Dear colleagues, I will. Uh... May I ask you to take your seats? Είστε παρακαλώ. May I ask you to take your seats? We would like to start the meeting. Καθίστε γιατί θα θέλαμε να αρχίσουμε και έχω πάρα πολλές ανακοινώσεις να κάνω. Έστω μεταξύ θα καταφτάσουν και οι συνάδελφοι. Λοιπόν, για την ημερήσια πρώτα απ' όλα. Ο εισηγητής ε, Δίας Δεμέρε για το σημείο 6 για το τριμερή διάλογο σε σχέση με τη Europol. Αυτό θα γίνει πριν το 5, ε, γύρω στις 10 παραδέταρτο. Εάν δεν έχετε αντιρρήσεις, εγκρίνεται η τροποποιημένη ημερήσια διάταξη. Στη συνέχεια έχω ολόκληρο κατάλογο ανακοινώσεων να κάνω για το γλωσσικό καθεστώς. Δεν έχουμε διερμηνία για τα ιστονικά, μαλτεζικά, σλοβενικά και ε, γαλλικιανά. Ζητούμε συγγνώμη. Στη συνέχεια πρέπει να εγκρίνουμε τις ε, συστάσεις των συντονιστών, κυρίως για το διορισμό ε, των ε, εισηγητών. Η κυρία Γκρίσβερ είναι η εισηγήτριά μας για την Συνεργασία Eurojust και Μαυροβούνη, κυρία Καόφμαν, σοσιαλιστές, εισηγήτρια για την εφαρμοστική απόφαση σε σχέση με τη Συμφωνία Συνεργασίας Eurojust και Ουκρανίας, ο κύριος Δεχόφσκι, ΕΛΚ, εισηγητής για την προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση για την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κυρία Μακόβη, συντηρητική εισηγήτρια για τις εγγνωμοδοτήσεις σε σχέση με τις εκθέσεις κόντ για την απαλλαγή 2014. Εγκρίνεται αυτές τις συστάσεις, νομίζω ναι. Θα πρέπει να ξέρετε ότι μια επιπρόσθετη συνεδρίαση θα γίνει στο Στρασβούργο στις 23 Νοεμβρίου. Θα πρέπει να ψηφίσουμε για τις ε, εκθέσεις οι οποίες έχουν αναβληθεί. Θα γίνει η ψηφοφορία τη Δευτέρα. Θα ψηφίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεση για τι συστάσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι διαπραγματεύσει για την Συμφωνία ΤΙΣΑ, για το εμπόριο σε υπηρεσίε Στη συνέχεια για τις ρυθμίσεις με την Ελβετική Συνομοσπονδία σε σχέση με τους όρους συμμετοχής της ε, στον ε, ΕΑΖΟ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υποστήριξη για το Άσυλο. Στη συνέχεια ειδική έκθεση για τον Ευρωπαϊκό Δημοσιολαβητή για την ε, έρευνα ιδίας πρωτοβουλίας για τον Frontex. Όλα αυτά θα γίνουν στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ τη Δευτέρα στο Στρασβούργο στις 23, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ας αρχίσουμε τώρα τη σημερινή μας συνεδρίαση. Μετά το πρώτο σημείο, γιατί προβλέπεται και η συζήτηση για τις ε, τρομοκρατικές επιθέσεις ε, στο Παρίσι θα ήθελα να τηρήσουμε ένα λεπτό σιγή ε, προς τιμή των θυμάτων. Ας γίνει αυτό πριν συζητηθεί ε, το θέμα. Τώρα θα συζητήσουμε τις τροπολογίες για την πρόταση για μια θεώρηση περιοδίας, σημείο 3. Ο κύριος Οχτωφέ, ο εισηγητής, θα πάρει τον λόγο πρώτος και μετά οι εισηγητές και μετά ενδεχομένως και η Προεδρία του Συμβουλίου, αν θέλουν να προσθέσουν κάτι. Κύριε Οχτωφέ, θέλετε να πάρετε τον λόγο. Oui, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που υπενθυμίζετε το επώδυνο περιβάλλον που προξένησαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις προηγουμένης Παρασκευής. Ευχαριστώ όλες τις χώρες και τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν εκφράζοντας τις, ε, τα συλληπιτήριά τους. Για την θεώρηση περιοδίας ε, που αναφέρατε, ε, βλέπω μια μορφή αγαθή αισιοδοξία, μακαρίου αισιοδοξία, που σχετίζεται με την υπόθεση αυτή και αναφέρομαι στη μεταναστευτική κρίση, αποκαλυπτική για την κοινή γνώμη των αδυναμιών μας, των αδυναμιών όλων μας, να προστατεύσουμε τι αδυναμίε όλων μας, να προστατεύσουμε τις χώρες μας την Ένωση από τις τρομοκρατικές επιθέσεις των οποίων η δικτύωση δεν σέβεται εθνικά σύνορα. Και έτσι βρίσκομαι εδώ ενώπιον σας ο συγητής ενός κειμένου που προτείνει τη χορήγηση θεωρήσεων σε κάθε υπήκο τρίτης χώρας με τρόπο που θα του επιτρέπει να κυκλοφορεί σε ολόκληρο το χώρο Σέγγεν για ένα έως και δύο έτη χωρίς βέβαια τη δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να περιορίζουν την κίνησή του, την κινητικότητά του και τις μετακινήσεις του στην επικρατεία τους. Είδατε και μια προηγούμενη εκδοχή του εγγράφου μου που προσπαθούσα να επανεστιάσω το πεδίο εφαρμογής σε πολύ συγκεκριμένες αλλά θεμητές κατηγορίες ε, υποψηφίων όπως είναι οι καλλιτέχνες, οι ε, υψηλών επιδόσεων αθλητές, το προσωπικό βέβαια που τους συνοδεύει, κατηγορίες για τις οποίες μπορεί, μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι είναι λογικό να γίνεται δεκτή η θεώρηση περιοδίας. Και τώρα προσπαθώ να επανεξισορροπήσω την ανάγκη να καλυφθούν ε, οι θεωρήσεις περιοδίας για τις κατηγορίες αυτές τις συγκεκριμένες και ταυτόχρονα διαφύλαξης ενός υψηλού επίπεδου ασφαλείας και ασφαλιστικών δικλείδων βεβαίως, ώστε να αποφύγουμε είτε τη στρέβλωση, είτε την καταστρατήγηση, είτε την απάτη. Και οι κύριες προτάσεις μου λοιπόν είναι οι εξής. Πρώτον, περιορισμός του πεδίου εφαρμογή για τους επαγγελματίες που έχουν θεμητό συμφέρον να κινούνται μέσα στο χώρο Σέγγεν για το πολύ μήνες. Για πάνω από τρεις μήνες. Δεύτερον, περιορισμός στο ένα έτος της διάρκειας αυτής της θεώρησης περιοδίας και τρίτον προσδιορισμός ορισμός κράτους αρμόδιου να εξετάσει την θεώρηση, το αίτημα θεώρησης με βάση το διάστημα της παραμονής στην επικράτειά του και όχι την πρώτη είσοδο του υποκειμένου της θεώρησης. Επίσης, μια διαδικασία πρώτερης διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών και την υποχρέωση ενημέρωσης για την παρουσία και ενδεχόμενο κίνδυνο για την ιστορική ασφάλεια του υποκειμένου της θεώρησης. Πέμπτο, κατάρτιση ενός πληρέστερου καταλόγου των δικαιολογητικών που θα χρειαστούν, θα χρειάζεται να ε, προσφέρονται να κατατίθενται, πάνω απ' όλα για να αποφύγουμε την στρέβλωση, την καταστρατήγηση ή την απάτη και βέβαια συνοδευτικά πληροφορίες ε, για άτομα γνωστά στις ε, προξενικές αρχές κτλ. Έκτον, σεβασμός των των δικαιοδοσιών των κρατών μελών. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή η θεώρηση περιοδίας να μετατραπεί σε μια μακροπρόθεσμη θεώρηση ε, μάλλον άδεια παραμονής και δεν μπορεί να δώσει δικαιώματα που αναγνωρίζει η άδεια παραμονή στα κράτη-μέλη. Πέραν αυτών των έξι προτάσεων έχουμε 57 τροπολογίες που κατατέθηκαν από, τους, από μένα, 72 δε από τους συναδέλφους στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Κάναμε συναντήσεις μεταξύ των ε, Σκιοδόνηση γητών και μου για να καταλήξουμε στα κύρια σημεία της προτάσεως που είναι όπως είπα ένα το πεδίο εφαρμογή, δύο η διάρκεια παραμονή στο χώρο Σέγγεν, τρίτον κριτήρια που προσδιορίζουν το αρμόδιο κράτος και τέταρτον ε, κατάλογος των δικαιολογητικών. Μπορούμε λοιπόν σε αυτό το στάδιο να διατυπώσουμε κάποια συμπεράσματα από τις ε, τροπολογίες που κατατέθηκαν ή αντίστροφα από αυτές που επελέγει να μην κατατεθούν. Πρώτον λοιπόν έχουμε να κάνουμε ένα κείμενο το οποίο αποκαλύπτει έως και αντιφατικές ή πάντως αποκλίνουσες προσεγγίσεις. Πρώτον λοιπόν έχουμε τους ε, βουλευτές που υπερασπίζονται την προσέγγιση της Επιτροπής. Αυτό τι σημαίνει συγκεκριμένα ότι προασπίζονται ένα άνοιγμα στο μέγιστο δυνατό αριθμό ετούντων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών. Και αυτό για μένα, ε, για μένα σημαίνει άπαντες όταν μιλάμε για τουρίστες. Εννοούμε τον κάθε Αυτό λοιπόν λέει η Επιτροπή, άνοιγμα και εξέταση του αιτήματο από το πρώτο κράτος εισόδου. Αντίστροφα, η πιο επιφυλακτική εναντί της προτάσεως Επιτροπής ε, ε, βουλευτές, αυτοί που ζητούν περιορισμό του πεδίου εφαρμογής και πιο αυστηρό ή πιο απαιτητικό κατάλογο δικαιολογητικών, γιατί έτσι μπορώ να εντοπίσω τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Πέραν αυτών των αποκλήσεων και πέραν αυτών των διαφορών, βλέπω ένα περιθώριο προόδου για να καταλήξουμε σε ένα ισορροπημένο κείμενο. Στην τεχνική συνάντηση που διεξήχθη εχθές μπορέσαμε να προχωρήσουμε σε, ως προς κάποιες διατάξεις, δηλαδή τη ε, διάρκεια της παραμονής <coughs> μέσα στο χώρο Σέγγεν μέχρι ενός έτους και τις αρχές που θα συμμετέχουν, ε, θα παρεμβαίνουν σε διαδικασίες. Ωστόσο και άλλες διατάξεις ακόμα βρίσκονται υπό συζήτηση και αυτές είναι το πεδίο εφαρμογή που για μένα έχει τεράστια σημασία γιατί προσδιορίζει το περιεχόμενο όλων των λοιπόν διατάξεων και άρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να περιλάβουν τους υπηκόους τρίτων κρατών ε, από τον κατάλογο του παραρτήματος 2 του κανονισμού 539 κάθετος 1, με χώρες όπως η Αλβανία ή η Μαλαισία, στην οποία σημειώνω πέντε άτομα υποψήφια για, ε, ε, ύποπτα για συμμετοχή στο ε, δίκτυο του Ισλαμικού κράτους και ενδεχομένως η διάπραξη τρομοκρατικών επιθέσεων στην Σύνοδο του ΑΣΕΑΝ ε, και άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν, θέλουμε, θέλω εγώ να δεχθώ την δυνατότητα συμπερίληψης ενός καταλόγου τόσο ευραίος ως κρατών ασφαλών προελεύσεων. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα βέβαια να χαιρετήσω την επικοδομητική στάση κατά την εξέταση των λοιπών άρθρων από τους συναδέλφους. Στα θέματα που ακόμα δεν έχουμε καταλήξει θα συναντηθούμε, θα συζητήσουμε και πάλι και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε, μια, σε ένα κείμενο ισορροπημένο που να την χάνει της υποστήριξη της πλειονότητας των συναδέλφων και πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λόπες Αργυγιάς, σκιώδης ηγητής για τους σοσιαλιστές δημοκράτες. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Φυσικά θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας εκφράζοντας τη βαθύτερη μου, τη βαθύτατη μου αλληλεγγύη προς τον γαλλικό λαό απέναντι στις φρικτές τρομοκρατικές ενέργειες που έγιναν στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου. Όλοι θα πρέπει να σταθούμε ως μια γροθιά ε, στο πλάι της γαλλικής δημοκρατίας, του γαλλικού λαού και βεβαίως γνωρίζω και συνειδητοποιώ την ευρωπαϊκή διάσταση αυτής της επίθεσης, αυτής της απόπειρας κατά τον πολιτισμό μας, των αξιών μας και φυσικά είμαστε έτοιμοι να συμφωνήσουμε στο γεγονός ότι αυτή η ρήτρα αλληλεγγύης ζήτησε ο πρόεδρος Ολάντ πριν από την επίσημη κοινή συνεδρίαση της ε, Εθνοσυνέλευσης και του Γερουσίας που καλεί ώστε να γίνουν βήματα από κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 47 της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, μας βρίσκει σύμφωνος. Τούτου λεχθέντος όλοι φυσικά ε, έχουμε Έχουμε όλοι μας ε, συμμετέχει σε συζητήσεις σε πολιτικού χαρακτήρα στις ομάδες μας τις τελευταίες μέρες. Φυσικά και ευχαριστώ τον κύριο Μπρίσορ για την εργασία του και για την παρουσίαση αλλά και για τις προσπάθειες που κατέβαλε ώστε να φτάσουμε σε κάποιο είδος συμβιβαστική, να βρούμε δηλαδή τρόπο ώστε να συνδυάσουμε τις θέσεις μας και να καταλήξουμε σε μία συνεπή ε, θέση του Κοινοβουλίου για την πρόταση περί της, ε, των θεωρήσεων περιοδίας. Έχω την ε, αναθεωρημένη εκδοχή του κώδικα θεωρήσεων και γνωρίζετε ήδη πως θελημένα απεφάσισα να μην καταθέσω τροπολογίες στην έκθεση αυτή καθώς συμμερίζομαι σε μεγάλο βαθμό την πρόταση της Κομισιόν δεν ε, ήθελα να καταθέσω τροπολογία σε μια πρόταση της Κομισιόν την οποία βρίσκω ε, ότι ε, αντιστοιχεί στο στόχο της. Προτιμώ να μείνω στην πρωτοβουλία της Κομισιόν. Στη διάρκεια της συνεδρίασης των συντονιστών, ωστόσο, είδαμε κάποιες απόπειρες για να μετακινηθούμε σε, σε έναν ευρύτερο, ευρύτερο ορισμό της θεώρησης περιοδίας και μέχρι στιγμής ε, προσπαθούμε να ε, ορίσουμε πολύ συγκεκριμένα το πεδίο εφαρμογή αυτή της πρότασης. Πέρα από τις ε, συνηθισμένες κατηγορίες, αθλητές, περιοδεύοντες καλλιτέχνε, θα μπορούσε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή ώστε να περιληφθούν και οι επιχειρηματίες ταξιδιώτε. Θα ήθελα επίσης να σκεφτούμε και κάποιες κατηγορίες τουριστών που θα μπορούσαν να ε, συμπεριληφθούν σε πεδίο εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλία, ώστε να συζητήσουμε και περαιτέρω αυτό το θέμα, ώστε να Ε, μπορέσουμε να βρούμε συγκεκριμένες θέσεις για τους ε, τουρίστες σε αυτό το φάκελο ε, που θα μπορούσε ενδεχομένω να διευρυνθεί στο μέλλον ανάλογα με το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Επίσης έχουμε προοδεύσει όσον αφορά τις αρχές, τον ορισμό των αρχών που συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες και στις ίδιες τις διαδικασίες γιατί έτσι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ η κυρία Βαλέρο. βάζεις και μικρό. Το μικρόφωνο είναι σβηστό. I pressed the wrong button. Λάθος κουμπί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει και θα ήθελα ε, να συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα για το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω αυτή την πρόταση και θα προτιμούσα την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κάποιες αλλαγές, μικρές αλλαγές που είχαμε προτείνει. τι έχουμε μπροστά μας. Έχουμε μια νομοθεσία η οποία θα ισχύει μακροπρόθεσμα και είναι συναισθηματικά φορτισμένοι λόγω της κατάστασης, ε, της χαοτικής ε, κατάστασης ε, με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, με τις επιθέσεις που έγιναν στο Παρίσι και προηγούμενες τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή συναισθηματικά να προσεγγίζουμε το ζήτημα, όμως ούτως άλλως συναισθηματικά φορτισμένο αυτό το θέμα και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ μιλώ με την ιδιότητα του νομομαθούς και θεωρώ ότι η νομοθεσία θα πρέπει να προβλέπετε για μακροπρόθεσμη εφαρμογή και επίσης μια νομοθεσία η οποία εύκολα θα μπορέσει να εφαρμοστεί από τις αρμόδιες αρχές. Θα ήθελα λοιπόν Ε, να υποστηρίξουμε την ε, πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι είναι πολύ περιοριστικές οι προτάσεις του εισηγητή και ε, διέπονται από συναισθηματικά επιχειρήματα και όχι ρεαλιστικά. Ευχαριστούμε κύριο Σκοράλ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι συμφωνώ όπως η κυρία Βαλέρο, ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ με την πρόταση της Επιτροπής είναι μια καλή και ισορροπημένη πρόταση σε σχέση με τους στόχους ε, της ε, διευκόλυνσης βέβαια και της κίνησης των ε, επισκεπτών καλλιτεχνών. Προφανώς οι τοποθετήσει του εισηγητή έχουν να κάνουν με τις τελευταίες επιθέσεις στο Παρίσι και είναι εύκολο να παρασυρθεί κανείς από τη συγκίνηση, όπω είπε και η Η πρόταση της Επιτροπής είναι αρκετά ισορροπημένη και την υποστηρίζουμε. Και πιστεύω ότι θα έπρεπε εκείνος ο οποίος θέλει να πάρει τουριστική θεώρηση να υπόκειται σε πιο πολλές απαιτήσει δικαιολογητικών από αυτές που αρχικά προβλέπονται. Όπως λέει και ο εισηγητής, βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει διευκόλυνση για καλλιτέχνες και λοιπό προσωπικό που ασχολείται στον χώρο του πολιτισμού, ανεξάρτητους επαγγελματίες και άλλους που θέλουν να μπορούν να παίρνουν από το ένα κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις για την εξασφάλιση δυνατότητα εργασίας και δεδομένου ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μερών ως προς την άδεια εργασίας, θα περιπλέκεται πάρα πολύ η κατάσταση εάν υπάρχει προϋπόθεση της άδεια εργασίας. Σε σχέση με τους καλλιτέχνες πρέπει να λάβουμε ιδιαίτερα την ε, διάσταση της μικρομισές επιχείρησης ε, με λογικές γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις ώστε να μην δυσκολεύεται ιδιαίτερα η δυνατότητά τους για περιοδία μέσα στην Ευρώπη. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τουριστική θεώρηση πρέπει να παραμείνει ε, ως το βασικό εργαλείο από 90 έως 120 ημέρες από 90 έως 180 ημέρες για τον ε, τουρίστα, περισσότερο για τον ε, καλλιτέχνη, ώστε να μπορεί να περιοδεύει για περισσότερο από 90 ημέρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. And I give now the floor to the Commission, please. Και τώρα το λόγο έχει η Κομισιόν. ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, τον εισηγητή καθώς και τους ευρωβουλευτές που πήραν το λόγο και που δίνουν τη στήριξή τους σε αυτήν το νέο είδος θεώρησης, αυτό πόσο το επανομαζόμενο ε, ε, την επανομαζόμενη μάλλον θεώρηση περιοδίας. Ε, η Κομισιόν ε, προτείνει μια, ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογής όχι για όλα τα άτομα τα οποία έχουν θεμητά ενδιαφέροντα να μείνουν στην στο χώρο Σέγγεν πάνω από 90 μέρες χωρίς να όμως να, μείνουν, να διαμείνουν σε κάποιο κράτος μέλος. Ακούσαμε τα σχόλια για περιορισμό του πεδίου εφαρμογής Πιστεύουμε πως ε, θα βρεθεί κάποια λογική συμβαστική σε αυτό. Θα είναι σημαντικό ωστόσο να μείνουν οι μεμονωμένοι ταξιδιώτες αλλά και αυτοί που δεν απαιτείται να έχουν βίζα ε, και που εν γέννη δεν αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ε, βεβαίωση για την σύνδεση με τις διμερείς που έχουν συλλάψει κάποια κρατημέλη με άλλες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να εκτιμάται η ε, αίτηση θεώρησης καθώς και το χρονικό διάστημα ισχύω της η Κομισιόν πρότεινε ένα χρόνο συν μια επέκταση του ενός χρόνου, παράταση. Ακούσαμε διάφορες προτάσεις. Αυτό θα μπορούσαμε φυσικά να το συζητήσουμε περαιτέρω σε σχέση με τα συνοδευτικά έγγραφα. Η πρόταση της Κομισιόν ήταν πολύ αυστηρή για αυτή την απέτηση, ότι δηλαδή ο ετών θα πρέπει να αποδείξει ότι πρέπει να μείνει πάνω από 90 μέρες σε κάθε κράτος μέλος και ότι έχει δυνατότητα ε, οικονομική για να παραμείνει για τη διάρκεια όλη αυτή τη χρονική Α Ας πούμε, μισθό ή, εν πάση περιπτώσει, αιτιολογικά, ε, δικαιολογητικά, ε, ώστε να, αποφύγουμε το κίνδυνο της ε, παράνομης μετανάστευσης. Το ίδιο ισχύει και ε, βέβαια για τα υπόλοιπα στοιχεία που ισχύουν και για το χώρο Σέγγιν, για τις συνηθισμένες θεωρήσεις δηλαδή, και αυτό ώστε να προλάβουμε τον κίνδυνο της παράνομης μετανάστευσης, αλλά και για να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας. Αυτά είναι λοιπόν τα σύντομα μου σχόλια από την πλευρά της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ από το πρόεδρο του Βίστον αν θέλει να παρέμβει. Όχι, δεν θέλει. γυρνάω στον ε, εισηγητή τότε, τον κύριο Ορτεφέ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους τους ε, συναδέλφους για τα σχόλιά τους και τις τοποθετήσεις τους. Όπως είπα και εισαγωγικά, έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Εγώ παραλαμβάνω τις επιφυλάξεις μας προς την πρόταση να συμπεριλαμβάνονται υπήκοοι τρίτων κρατών που δεν ε, λαμβάνουν θεώρηση για συγκεκριμένο στόχο και για τους οποίους θα είναι πολύ δύσκολο να διαγνωστεί η πορεία και η περιοδία μέσα στην Ένωση. Ε, πάντως είπα και νωρίτερα ότι θεωρώ πως υπάρχει περιθώριο ε, προόδου και θα συνεχίσω προς αυτήν την κατεύθυνση να εργάζομαι ε, μια νέα συνάντηση μεταξύ ε, σκιωδών εισηγητών προβλέπεται για την επόμενη εβδομάδα και βεβαίως θα προσπαθήσω να ε, προωθήσω λύσεις συμβαστικές, πρόοδο και βέβαια στο δυνατόν ταχύτερα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ορτεφέ και περνάμε στο άλλο θέμα που έχει να κάνει με τη θεώρηση των διαβατηρίων με τον κύριο Λόμπες Αγγιλιάρ για, τις, ε, για τον ε, κώδικα της Ένωσης για τη θεώρηση διαβατηρίων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και πάλι. Θα ήθελα να κάνω κάποια γενικά σχόλια. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και τους σκιώδεις εισηγητές για τις τροπολογίες που υπέβαλαν. Σημείωσα τις θέσεις τους και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή με τους σκιώδεις εισηγητές να καταλήξουμε συμβαστικές τροπολογίες που θα ενσωματώνουν στο δυνατόν περισσότερες τροπολογίες είναι δυνατόν. Είναι ζωτική σημασία να έχουμε μια στενή συνεργασία ώστε να είναι πάρα πολύ καλή η διαπραγματευτική θέση της Επιτροπής μας εν και των μελλοντικών διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Θα πρέπει να δράσουμε με στρατηγικό τρόπο, να έχουμε κατά νου πάντοτε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Όσες φορές χρειαστεί θα συναντηθώ με τους σκιώδεις εισηγητές στις ε, συσκέψεις που διοργανώνουμε ή και διμερώς. Είμαι στη διάθεσή σας. Έχουμε δουλειά μπροστά μας. Έχουμε αρκετές τροπολογίες. ...357 συγκεκριμένα. Είναι η πρώτη και σίγουρα όχι η τελευταία συνεδρίαση για την εξέταση των τροπολογίων δηλαδή. Έχουμε ήδη κάνει τρεις ε, σκέψεις σκιωδών και την επόμενη εβδομάδα θα ξανασυναντηθούμε στο Στρασβούργο για να δούμε πώς θα έχει το θεμα... το... η μερίσια διάταξη, το χρονοδιάγραμμα μάλλον. Θέλουμε το αργότερο να ψηφίσουμε μέχρι το πέρας του τρέχοντος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με την επόμενη Προεδρία, την Ολλανδική, για τις ε, τροπολογίες. Υποστηρίζω την ιδέα της διευκόλυνσης ε, που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτός είναι ο στόχος. Διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων ε, διότι είναι επαχθείς και χρονοβόρες τώρα οι διαδικασίες βάσει του ισχύοντος κανονισμού. Γι' αυτό και τροποποιούμε τον κανονισμό για να διευκολύνουμε ναι. ε, την ε, έκδοση θεωρήσεων, ούτως ώστε με ένα απλούστερο νομικό πλαίσιο να μπορούν να ταξιδεύουν ευκολότερα οι άνθρωποι. Υποστηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής και τις τροπολογίες που ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση, διευκόλυνση. Κυρίως για ευραχίδες. Μετά από κάποια χρόνια εφαρμογής βλέπουμε πόσο επαχθείς είναι οι διαδικασίες. Επίσης έχουμε ε, συντομότερες ε, προθεσμίες ε, κατάλογο ταξιδιωτών VIS υποχρεωτική εκπροσώπηση εκπροσώπηση, προσδιορισμός των στενών συγγενικών προσώπων, θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων. αυτά είναι τα βασικά σημεία της τροποποιητικής ε, νομοτεχνικής διαδικασίας. Έχουμε υψηλότερες, υψηλότερα τέλη για τις θεωρήσεις σε κάποιες τροπολογίες. Ας ε, επιδιώξουμε έναν εξορθολογισμό των τελών. Δεν θα πρέπει να είναι αποτρεπτικά υψηλά τα τέλη. Ε, όσοι έχουν το νομικό δικαίωμα να μετακινηθούν δεν θα πρέπει να προσκρούν σε αυτό το εμπόδιο. Επίσης μιλήσαμε για την ταξιδιωτική ιατρική ασφάλεια, όμως τη διέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της. Θα συμφωνήσω. Οι τροπολογίες του ΕΛΚΑ και των συντηρητικών θέλουν να επανεισάγουν την υποχρέωση υποχρεωτικής ταξιδιωτικής ασφάλειας. Θα ήθελα να διευκρινίσει και πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόθεσή της. Γιατί διέγραψε την ε, ιατρική ε, υποχρεωτική ασφάλεια. Για να έχουμε περισσότερα στοιχεία, για να αναλύσουμε το θέμα, θα είναι σημαντικό αυτό για τις διαπραγματεύσεις μας και για τη θεώρηση περιοδίας. Υπενθυμίζω πως η ιατρική ταξιδιωτική ασφάλεια δεν είναι όρος εισόδου ε, βάσει του τωρινού τελωνιακού κώδικα Σέγγεν, δεν συνιστά ε, προϋπόθεση γιατί λοιπόν θα πρέπει να ε, αποτελεί όρο για τον κώδικα των θεωρήσεων. Θα πρέπει να υπάρχει και συνέπεια, συνοχή ανάμεσα στα δύο. Θα ήθελε να μας το διευκρινίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τις τροπολογίες που σχετίζονται με τον ορισμό των στενών συγγενικών προσώπων. Απευθύνω έκκληση για την υποστήριξη της θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεωρώ πως η σωστή προσέγγιση θα ήταν να υποστηρίξουμε το στόχο διευκόλυνση έκδοσης οικογενειακών θεωρήσεων για την υποχρεωτική εκπροσώπηση θα συμφωνήσω με του συναδέλφου με τι τροπολογίε που υποστήριξαν την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη τελευταία συνάντηση των σκιωδών ε, αποφασίσαμε να κάνουμε κι άλλο ένα βήμα προ αυτή την κατεύθυνση, ακολουθώντα διατύπωση Επιτροπή Τραν. Δηλαδή, στοιχείο γεωγραφική, το στοιχείο τη γεωγραφική απόστασης μέχρι το προξενείο, καθώς και ε, το χρόνο μετακίνησης. Πόσο η ώρα πόσο χρόνο ε, θα διαρκέσει το ταξίδι. Επίσης, ε, κανονικοί, τακτικοί ε, ταξιδιώτες VIS. Έχω καταθέσει και συμβαστική τροπολογία για αυτό το ζήτημα. Ελπίζω να εγκριθεί. Βασίζομαι στην εξή λογική. Προσπαθώ να ικανοποιήσω τα αιτήματα του ΕΛΚ και ε, τρεις είναι οι που απαιτούνται τώρα για να θεωρηθεί κάποιος ε, συνήθις ε, τακτικός ε, ταξιδιώτης. Νομίζω ότι πρέπει να παρατείνουμε το χρόνο για την ε, έκδοση αυτών των θεωρήσεων. Δηλαδή, αν κάποιος έχει θεώρηση πολλαπλών θεωρήσει αυτός ή αυτή ως τακτικός ταξιδιώτης. Αυτή είναι η... Ε, αυτό η αυτο ειναι το σκεπτικό. Όμως πρέπει με νόμιμο τρόπο, με νόμιμο τρόπο να έχουν χρησιμοποιηθεί αυτές οι θεωρήσεις. Δεν μπορούμε όμως να διαφοροποιούμε ανάμεσα σε επικούς ε, τρίτων χωρών και υπηκός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε? τρίτων χωρών όπως βλέπουμε σε μια τροπολογία. Διάβασα ε, τροπολογίες που ακολουθούν αντίθετη κατεύθυνση. Εγώ προσπαθώ με τους σκιώδες να καλύψω τα αιτήματα όλων των ε, πολιτικών ομάδων. Γιατί η νόμιμη εκπροσώπηση ε, χρειάζεται για κάποιους που ταξιδεύουν σε μακρινές αποστάσεις για να μπορέσουν να καταθέσουν ε, καν ε, την αίτηση, να πάνε στην πρωτεύουσα και στο προξενείο το αρμόδιο για να μπορέσουν να ζητήσουν τη θεώρηση. Καλό θα ήταν αν ε, υπάρχουν προξενία σε άλλες γειτονικές χώρες να έχουν τη δυνατότητα και εκεί να υποβάλουν την αίτηση θεώρησης. Γι' αυτό και κατέθεσα την αντίστοιχη τροπολογία για να διευκολύνουμε ε, υπό ορισμένε ε, συνθήκες ε, την έκδοση θεωρήσεων και σε άλλα προξενία. Τροπολογία 15. Ναι, ναι, ένα λεπτάκι. Υπάρχει και το πάρα πολύ σημαντικό θέμα των ανθρωπιστικών θεωρήσεων. Το ξέρουν οι συνάδελφοι ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα διότι είναι μια ευκαιρία για να ενισχύσουμε το δυναμικό των ανθρωπιστικών θεωρήσεων υπάρχουν ανακολουθίες στον τωρινό κώδικα θεωρήσεων. Τα άρθρα 19 και 25 είναι αντιφατικά. Στον τωρινό κώδικα, στο 19 δεχόμαστε τις προϋποθέσεις και στο 25 παραπέμπουμε στον κώδικα Σέγγεν. Θα πρέπει να διευρύνουμε τις νόμιμες οδούς εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν υπάρχουν αυτές, ε, τι μπορεί κάποιος να κάνει παράνομα να προσπαθήσει να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταφύγει σε ε, διακινητές ε, και έτσι από τη μετανάστευση την νόμιμη μετανάστευση περνάμε στην παράνομη μετανάστευση και καταλήγουμε στο χάος που έχουμε τώρα με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα συμφωνούν μαζί μου. Εγώ υποστηρίζω το 309 για την θέσπιση μιας ανθρωπιστική θεώρησης και ε, για ένα συνεκτικό πλαίσιο σε σχέση με τα πολλά διαφορετικά καθεστώτα που ισχύουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα μέσα που τώρα είναι διαθέσιμα για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις στην αναθεωρημένη εκδοχή του κανονισμού θα πρέπει να ασχοληθούμε αυτό το ζήτημα είναι στον πυρήνα αυτής της ανθρώπινης τραγωδίας. Είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε διευκνήσεις και σας ευχαριστώ για την προσοχή που δείξατε. Ναι, έχουμε πολύ λίγο χρόνο πια. Παρακαλώ, ποιος αντικαθιστά τον κύριο Μπέκερ. Ναι, πρόεδρε, ο κύριος Οχτεφέ, εκ μέρους του συνάδελφου Ντεμπάκερ, δεν μπορούσε να παρών. Προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε συμβαστικές ε, λύσεις, ε, οι συζητήσεις συνεχίζονται, πρόκειται να γίνει συζήτηση την επόμενη εβδομάδα και κάποιες λύσεις ακόμη δεν είναι μεν ικανοποιητικέ. Ελπίζουμε ωστόσο να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση. Για το ΕΛΚ σημασία έχει να διατηρήσουμε ένα περιθώριο χειρισμών έτσι ώστε εν τέλει να ε, υλοποιηθούν αυτές οι προτάσεις. Θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στην τροπολογία 195 των συνάδελφων ε, Hans Becker και του υποφαινομένου που στόχο έχει την τροποποίηση του άρθρου 21 παράγραφος 3 όπου η πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει θεώρηση τριών ετών με πολλαπλές εισόδους για αναγνωρισμένους και καταγεγραμμένους στο σύστημα του Σέγγεν ταξιδιώτες που ήδη έχουν κάνει νόμιμη χρήση της θεώρησής τους. Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πρέπει αυτός ο όρος να αντικατασταθεί, το χορηγείται, από το δύναται να χορηγηθεί στην ε, πρόταση. Δηλαδή για μας κάποιος ο οποίος έχει επανειλημμένος χρησιμοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο το δικαίωμα της θεώρησης, κατά κανόνα δεν πρέπει να αποκλείεται, αλλά δυστυχώς υπάρχουν εξαιρέσεις και άρα πρέπει τα προξενία να έχουν ένα περιθώριο δράσος, να μπορούν να αντιδρούν, να ε, αρνηθούν ακόμη τη χορήγηση της θεώρησης εάν ε, υπάρχει λόγος να ε, απορριφθεί το αίτημα. Και επίσης υπάρχουν και άλλες πτυχές, αγαπητή συνάδελφοι κυρία Πρόεδρε, το ζήτημα της, ασθε... της ασφάλισης το άρθρο 33 για τις ε, θεωρήσεις ε, σε άτομα που υπόκεινται σε προσωρινό καθεστώς. Ε, όλα αυτά πρέπει να γίνουν δεκτά και εκ μέρους του συναδελφού Χατσπέκερ θα ήθελα να εκφράσω ευχαριστίες για το πνεύμα συμβιβασμού το οποίο επιδείξατε. Ευχαριστώ Βαλερό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πολύ καλή δουλειά κάνει. Όντω είναι καλή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, συμφωνώ και με τις προτάσεις που κατέθεσε ο εισηγητής. 357 ε, ε, τροπολογίες έχουμε για το τροποποιημένο κώδικα θεωρήσεων και αυτό δείχνει πόσο μεγάλο ενδιαφέρον, πόσο ε, μεγάλο ειδικό βάρος πιστεύουν όλοι οι βουλευτές ότι έχει η τροποποίηση αυτού του κανονισμού. Θεωρούμε ότι πρέπει, όπως και στο προηγούμενο θέμα, να μπορέσει να ισχύσει μακροπρόθεσμα η νέα νομοθεσία και να μην δημιουργήσει περισσότερο μεγαλύτερο χάος όπως αυτό που βιώνουμε τώρα με τις επιθέσεις και την προσφυγική χρήση. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με τη διατύπωση. Το σημαντικό είναι ότι μιλάμε για τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης και η Επιτροπή ή ακόμη και το Συμβούλιο μιλάει πλέον για νόμιμες οδούς μετανάστευσης. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπίσουμε αυτές τις νόμιμες οδούς και ε, να υποστηρίξουμε και τις προτάσεις για την ανθρωπιστική θεώρηση. Το χρειαζόμαστε για να σώσουμε ζωές πλέον στη Μεσόγειο. Επίσης ε, θεωρώ ότι το τέλος για τις ε, ε, θεωρήσεις ε, ορισμένες φορές είναι υπερβολικά υψηλό, κυρίως για ανθρώπους που έρχονται από χώρες χαμηλού εισοδήματος. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε με τον εισηγητή ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστούμε ο κύριος Κοράου. Παρακαλώ σύντομα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θα προσπαθήσω. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά του. Η προσέγγιση είναι θετική, την υποστηρίζουμε και ιδιαίτερα στη δυνατότητα χρήσης, ε, σε, εξασφάλιση πολύ στο χρονικό διάστημα θεώρηση Σέγγεν για ανθρωπιστικούς λόγους και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που χρειάζονται άσυλο. Πρέπει να φτάνουν στην Ευρώπη πολύ σύντομα και χωρίς περιπλοκές. Κάνουμε τροπολογίες που συμπληρώνουν, δεν επαναλαμβάνουν το έργο του εισηγητή, ιδιαίτερα σε σχέση με την προσθήκη στο άρθρο 2, ανάγκη για προσθήκη, προσθήκη μιας αναφοράς στους ανθρωπιστικούς λόγους που θα εξασφαλίσουν μια παρέκκληση για την δυνατότητα χορήγησης θεώρησης για λόγους ανθρωπιστικούς. Η 137 επίσης καλύπτει το ίδιο ε, την ίδια στόχευση. Κάτι άλλο που δεν καλύπτει επαρκώς ε, η πρόταση της Επιτροπής είναι αυτό το σχετικό με τα άρθρο 10 και 19, με το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι δεν χρειάζεται τόση πολύ εστίαση στο κίνδυνο από τη, από τη λαθρομετανάστευση νομίζω ότι θα πρέπει άπαξ και περάσουν οι προθεσμίες αναφέρει ο εισηγητής να καταπίπτει η δυνατότητα για τη θεώρηση. Αυτό όμως ε, θέτει ένα ιδιαίτερο βάρος και ε, υπο, καχυποψία εις βάρος ε, των ετούντων και βεβαίως των ιδίων και των οικογενειών τους σε περίπτωση παρα, παραμονής μεγαλύτερης από την υποχρεωτική διάρκεια της θεώρησης. Επίσης νομίζω ότι θα πρέπει σε περίπτωση που γυρινοποίηση των διαδικασιών με βάση τον κώδικα να είναι αυτές πιο αυτοματοποιημένες, λιγότερο γραφειοκρατικές και να επιτρέπουν τη χορήγηση της θεώρησης σχετικά γρήγορα στον ετών. Ευχαριστώ κυρία Βεργία. Σύντομα. Ναι, θα είμαι σύντομη. Θα ήθελα καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Ορτοφέ γιατί δεν ήμουν παρούσα για την προηγούμενη συζήτηση, αλλά ταυτόχρονα εργαζόμαστε για αυτές τις δύο εκθέσεις και η λογική της ομάδας μου είναι η ίδια και για τα δύο κείμενα. Θα εστιάσω ωστόσο τώρα στην έκθεση του κυρίου Αγγιλάρ. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε δεδομένου του σημερινού πλαισίου τον αρχικό στόχο αυτής της αναθεώρησης που στόχο είχε να διευκολύνει τη ζωή ανθρώπων που τακτικά ε, μεταβαίνουν για επαγγελματικούς λόγους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την εντύπωση ότι ε, υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με την Κομισιόν που δεν ανησυχεί τόσο για τα θέματα ασφάλειας και βρίσκω ότι αυτό είναι κρίμα. να θυμίσουμε τα εξή. Δεν θα πρέπει αυτή η αναθεώρηση να αμφισβητήσει κάποιες αρχές που οδηγούν, καθοδηγούν τις ενέργειες της Ένωσης στον τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά το ε, δικαίωμα για ε, οικογενειακή επανένωση και επίσης όσον αφορά το δικαίωμα στην υγεία. Γιατί υπάρχουν κάποια σημεία που δημιουργούν πρόβλημα. Αλλά ελπίζω τουλάχιστον να βρεθεί μια λύση. Για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις επίσης να θέλω να πω δύο λόγια, γιατί ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουμε προβλήματα στα ευρωπαϊκά σύνορα ακριβώς οφείλεται στο ότι αυτοί οι πρόσφυγες δεν καταφέρνουν να ζητήσουν το άσυλο υπό μαλές συνθήκες. Όταν βλέπω ότι τα όσα προβλέπει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Άνοιξη έχουν επιτρέψει μόνο σε 150.000 ε, ε, ανθρώπους να μπουν στην Ένωση, λέω ότι στην ουσία κάνουμε βήμα σημειωτών και πρέπει κάτι να αλλάξει σε αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βερζιά. Θα στραφώ τώρα στην κυρία ε, Καρζία γράφω. Σύντομα παρακαλώ. Μάλιστα, Πρόεδρε, για αυτά που αναφέρθηκαν για την ασφάλιση ε, η Κομισιόν δεν έχει επαρκείς ε, αποδείξεις για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής ασφάλισης. Δεν είναι απέτηση και ούτε ελέγχεται ε, στα σύνορα. Έχουν υπάρξει τέτοιες καταγγελίες για απλήρωτους νοσοκομιακούς λογαριασμούς, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ακόμα σαφές κατά πόσο αυτοί οι λογαριασμοί αντιστοιχούν σε πολίτες τρίτων χωρών που υποχρεούνται σε θεώρηση ή όχι, ή ακόμα και σε Ευρωπαίους πολίτες για το θέμα της διευκόλυνσης για στενούς συγγενεί Ευρωπαίων ε, πολιτών θέλαμε να τον εναρμονίσουμε αυτό για τους ε, ε, συγγενείς, στενούς συγγενείς, οικογένεια, αλλά και για τους πολίτες που έχουν ασκήσει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας αλλά και αυτούς που δεν το έχουν ασκήσει, να υπάρχει εναρμονισμένη δηλαδή προσέγγιση. Για τους τακτικούς ταξιδιώτες υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε σχέση με το όριο, το τι σημαίνει συχνός ταξιδιώτης. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες διευκολύνσεις και τις προσφέρουμε αυτούς, ε, αυτές για τους ε, ε, ταξιδιώτες ε, καλής πίστης. Συμμεριζόμαστε την αρχή όσον αφορά τι νόμιμε οδού μετάβαση στην Ένωση, αλλά πιστεύουμε πως αυτό δεν είναι το σωστό νομικό μέσο, διότι αναφέρεται μόνο σε θεωρήσεις μικρής ε, διάρκειας. Αλλού θα πρέπει αυτό να ρυθμιστεί και αυτά είναι τα σχόλιά μου. Σα ευχαριστώ πολύ. Η Προεδρία του Λουξεμβούργου θέλει να παρέμβει. Να είστε Σύντομοι. Κύριε Πρόεδρε, εξότιμοι κυρίε και κύριοι, βουλευτές. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Σε σχέση με την ανάλυση από πλευράς της Επιτροπής της αναδιατύπωσης του κώδικα αλλά των θεωρήσεων αλλά και των θεωρήσεων περιοδίας βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιταχυμένη διαδικασία. Κάποια άρθρα όμως ζητήθηκε από το Τζάι του Οκτωβρίου να ξανασυζητηθούν. Με επιφύλαξη λοιπόν και ανάλογα με τις εξελίξεις στο Τζάι θα προχωρήσουμε της εργασίας μας ως Προεδρία μέχρι το τέλος του 2015. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η αναδιατύπωση του κώδικα θεώρησης σημαίνει για το Κοινοβούλιο, για το Συμβούλιο, ε, εξέταση μόνο των προτάσεων από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ο εισηγητής, ευχαριστώ πολύ και ιδιαίτερος για την υποστήριξη που εκφράζεται στις θέσεις του εισηγητή σας. Ε, καθώς και την διάθεση για συμβιβασμό από πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η διευκρινής Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την ε, δυσκολία προσδιορισμού της απέτησης για την ιατρική, των όρων δηλαδή, της των όρων ε, για την ιατρική θεώρηση. Είναι δύσκολο να διαγνωστεί αυτό, αλλά το να περιοριστούμε μόνο σε μονογραφικές θεωρήσεις. Γιατί εγώ θα ήθελα να ανοίξει αυτή η νόμιμη οδός προς όλους εκείνους που θα ήθελαν νόμιμα και για λόγους ανθρωπιστικούς ε, θα είχαν ανάγκη να μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει βεβαίως ε, να κοιτάξουμε κάθε διαφορετική περίσταση και περίπτωση. Καλώς λέει η Πρόεδρος, 10... Ε, για τις 30 Νοεμβρίου έχει προβλεφθεί η ψηφοφορία. Το επόμενο θέμα μας είναι η έκθεση υπεπραγμένων από τον τριμερή διάλογο για τη Europol και έχετε το λόγο κύριε Δίας Δεμέιρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου με τον ε, γαλλικό λαό και με τις ε, αρχές, τις γαλλικές αρχές ε, ενώπιον της τραγωδίας. Θέλω επίσης να εκφράσω την αποφασιστικότητά μου, την ευθύνη μου, την ευθύνη που νιώθω ως νομοθέτης και που θα πρέπει να αποδειχτεί μέσα σε ένα λεπτό. Ε, κοινοβούλιο και Europol. Ενημερωτικά, ε, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι έχουμε κάνει εννέα τριμερείς διαλόγους, τρεις ε, υπό την Ιταλική Προεδρία, τρεις υπό τη Λετωνική Προεδρία και τρεις ε, υπό την σημερινή Προεδρία του Λουξεμβούργου. Επιπλέον έγιναν 10 τεχνικής φύση συνεδριάσεις. Ο επόμενος τριμερής διάλογος και μάλλον ο τελευταίος ή άντε ο προτελευταίος θα γίνει την επόμενη 5η 26 Νοεμβρίου. Στη διάρκεια του περασμένου τριμερούς και με βάση κάποιες συμβιβαστικές που είχα προετοιμάσει προσπαθήσαμε να συμφωνήσουμε επί τριών θεμάτων που εξακολουθούν να είναι ανοιχτά αλλά που έχουμε πολλές πιθανότητες να τα κλείσουμε σε, με πολύ ψηλό επίπεδο συνένεσης και μιλώ για το κοινή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου στην ε, υποψηφιότητα του εκτελεστικού διευθυντή στη συνεργασία των ε, υφιστάμενων δομών για τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Ήρου, την ε, μονάδα περιεχομένου στο ίντερνετ και οι πληροφορίες, η μονάδα για τις πληροφορίες ιδιωτικού χαρακτήρα. Φτάσαμε λοιπόν στην συνένεση ότι μια μικρή ομάδα σύνταξης θα συντάξει συμβιβαστικές λύσεις και θα μας τι στείλει ώστε να εξετάσουμε κατά πόσο συμφωνούμε ή όχι. Αυτό μάλλον θα γίνει στη διάρκεια της ε, σήμερων. Οπότε το μόνο θέμα που παραμένει ανοιχτό είναι αυτό που, αφορά το Ήρου, ε, δηλαδή εκείνη την μονάδα για το περιεχόμενο του ίντερνετ και περιμένουμε ε, πολύ θετικές ε, αντιδράσεις ώστε να δώσουμε πηγόντως απάντηση όσον αφορά και μάλλον υπογραμμίζω την λέξη πήγων ιδιαίτερα απέναντι στην τρομοκρατική απειλή. Εννοείται ότι πρωταρχική αξία είναι η ασφάλεια των συμπολιτών μας σε μια δημοκρατική και ελεύθερη κοινωνία, όπως, όπου οι αρχές ασφαλείας των κρατών και των αντίστοιχων αρμόδιων μάλλον αρχών της Europol συγκεκριμένα για τα θέματα ασφάλειας, θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να μπορούν επιγόντως να προλαμβάνουν αλλά και να καταστέλουν τις τρομοκρατικές ενέργειες που μας ε, ε, απειλούν και που μας ε, βλάπτουν. Ο εισηγητής και η ομάδα του λοιπόν στηρίζουν μία ενιαία νομοθετική πράξη και μάλιστα με σύμφωνη και επίγουσα μεταγραφή και εμείς εκτιμούμε την προσπάθεια των σκιωδών για την επίτευξη αυτού του στόχου. Πάντως σε κάθε περίπτωση και με μεγάλη ταπεινοφροσύνη θα ήθελα να πω ότι αν οι, βοήθειές, οι προσπάθειές μου δεν ευοδοθούν, παραμένω ε, αποφασισμένος ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε, διότι ο τρόμος δεν ξεκουράζεται ποτέ. Όπως ε, δείχνει άλλωστε και η εξάρθρωση χθεσινή του, της κλίκας του Σεντενή που ήταν έτοιμη και, και, και που προετοίμαζε επιθέσεις ε, στο αεροδρόμιο Σαρντεγκολ και στο οικονομικό κέντρο του Παρισιού. Και εγώ ζητώ λοιπόν να ε, μπορέσουμε να ενεργοποιηθούμε και να καταπολεμήσουμε αυτήν την ε, θανατηφόρα πληγή. Δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα, είναι θέμα ρεαλισμού, ε, να έχουμε ένα ρεαλιστικό όραμα για το ποια είναι η ευθύνη μας ως νομοθέτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Δίας Δεμέρα. Και τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως όλοι γνωρίζουμε, την περασμένη Παρασκευή το βράδυ έγινε στο Παρίσι φοβερές μάλλον τρομοκρατικές επιθέσεις με θύματα 130 ανθρώπους. Η Γαλλία ε, ε, ε, κήρυξε τριήμερο πένθος και για μας σε ολόκληρη την Ευρώπη τηρήθηκαν ε, λεπτού, ενός λεπτού σιγής. Όπως ξέρετε εμείς ακυρώσαμε την περασμένη Δευτέρα τη συνεδρίασή μας για να επιτρέψουμε μια περίοδο πένθους και προβληματισμού πριν έρθουμε στις συνεδριάσεις μας. Όλοι μας συγκλονιστήκαμε από αυτές τις φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις που σκότωσαν και πλήγωσαν ένα σωρό κόσμο και οι σκέψεις μας ε, βρίσκονται κοντά στα θύματα και τις οικογένειές τους. Θέλω να, να διαβεβαιώσω τους Γάλλους συναδέλφους για την βαθιά μας αλληλεγγύη και θα ήθελα να σας καλέσω να τιμήσουμε τα θύματα τηρώντας ενός λεπτού σιγή. Παρακαλώ. now debate. It is the duty of our committee. Συνεχίζουμε για την καθήκον της Επιτροπής μας των Ευρωπαϊκών Θεσμών και των κρατών μελών στο σύνολό τους είναι να θεσπίσουν τα απαραίτητα μέσα και τις λειτουργικούς πόρους για να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία. Η Ευρώπη είναι ενωμένη στον αγώνα κατά του της τρομοκρατίας και είναι αποφασισμένη να εντοπίσει τα δίκτυα και όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση αυτής της ε, δεχθούς πράξης. Αυτή είναι η δέσμευσή μας και τώρα πρέπει να επιταχύνουμε τις εργασίες μας για αυτό το θέμα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Όπως γνωρίζετε, μια, ένα έκτακτο συμβούλιο, ε, έκτακτο εσωτερικών υποθέσεων και δικαιοσύνης έχει διοργανωθεί για τις 4 αύριο το μεσημέρι και είμαι ευτυχή που οι βασικοί συμμετέχοντες ε, θα είναι εδώ για να μας ε, ενημερώσουν για το τι θα γίνει και Θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο και να καλωσορίσω εδώ τον ε, πρέσβη Μπράουν που αντιπροσωπεύει την Προεδρία του Συμβουλίου και που σύντομα θα μας εκθέσει τα όσα θα συζητηθούν στην έκτακτη σύσκεψη του Συμβουλίου Τζάι αύριο και τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Στη συνέχεια θα δώσω συντομία το λόγο στον άλλο μας προσκεκλημένο που αντιπροσωπεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Βέτερ. Και τέλος θα ακούσουμε τον κύριο Βιμ από την ε, διάθεση της Europol που θα εκθέσει στους ευρωβουλευτές την προοπτική ε, και την απάντηση που μπορεί να δοθεί σε, αυτές, σε αυτά τα γεγονότα. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο σε εσά ε, για σχόλια. Πρώτα λοιπόν η Προεδρία του Συμβουλίου κύριε Μπράουν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μετά τα τραγικά περιστατικά της ε, Παρασκευής και τους νέους συναγερμούς, εχθές και προχθές, θεώρησα απαραίτητο να γίνει μια έκτακτη συνεδρία των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνη, ώστε να καταγράψουμε τι τελευταίε εξελίξει. Τα γεγονότα, αλλά και την ανταπόκριση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα γεγονότα και τον τρομοκρατικό κίνδυνο. Την απειλή αυτή που είναι πραγματική και που υλοποιήθηκε κατά τρόπο τραγικό. τι Κυριακή λοιπόν, σε συνεννόηση με τις γαλλικές αρχές αποφάσισε η Λουξεμβουριανή Προεδρία να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση για την Παρασκευή αύριο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, ειδικά αφιερωμένη σε άμεση απάντηση σε ζητήματα, όχι δηλαδή μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μιας στρατηγικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά άμεσες απαντήσεις. υπόθηκε βεβαίως ότι η ανταλλαγή πληροφοριών δεν ήταν ή ενδεδειγμένη ή ότι κάποια μέτρα θα έπρεπε να ληφθούν την επαύριο των αποφάσεων που ακολούθησαν τις επιθέσεις Αρλή και που δεν υλοποιήθηκαν εν τέλει. Όλα αυτά μας οδηγούν σε επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί και την υπογράμμιση νέων στοιχείων έμφασης στην καταπολέμηση τρομοκρατίας και ίσως και ο διευθυντής της Europol να επανέλθει στο θέμα αυτό. Ιδιαίτερα θέματα ανταλλαγής πληροφοριών στα οποία εγώ δεν θα σταθώ. Έχουμε λοιπόν εμείς οι Υπουργοί ένα σχέδιο συμπερασμάτων για το Συμβούλιο λειτουργικού χαρακτήρα, επιμελητιακού χαρακτήρα, όχι δηλαδή ε, γενικής πολιτικής, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ιδιαίτερα για την αναθεώρηση στρατηγικής γιατί θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό αργότερα. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Σύστημα Πληροφοριών ε, για τα προσωπικά δεδομένα, ο έλεγχος των, ε, του εμπορίου ε, πυροβόλων όπλων, ανταλλαγή συστηματική πληροφοριών, συστηματική έλεγχη και ενισχυμένη έλεγχη στα σύνορα σε σχέση με τις ε, τρομοκρατικές ροές, επέκταση της εφαρμογής του συστήματος τίκρης που είναι το ποινικό μητρό για επικόους τρίτων κρατών και πολύ σύντομα Βλέπετε λοιπόν ότι είναι απαραίτητο στα μάτια του Συμβουλίου να προχωρήσουμε ταχύτατα στην υπόθεση αυτή. στα θέματα αυτά που είναι δύσκολα, που είναι απαραίτητο να εξεταστούν και που έχουν να κάνουν βέβαια και με τον περιορισμό τόσο των αδικημάτων όσο και των στοιχείων που έχουν να κάνουν με την διάρκεια διατήρησης δεδομένων, διακράτηση δεδομένων. Δεν ήρθαμε για να διαπραγματευτούμε το θέμα αυτό, γίνεται η διαπραγμάτευση. Οι Υπουργοί θα καταγράψουν και θα προσπαθήσουν να δώσουν τα στοιχεία δυναμικής που απαιτούνται στη διαδικασία αυτή προκειμένου να χαλαρώσει κατά κάποιον τρόπο, να καταστεί πιο ήπια η περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται. Για τον έλεγχο των όπλων. Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρετε, πρέπει να χαιρετήσουμε την οθέτηση, μια απόφαση για την υλοποίηση της συμφωνίας για την διάθεση όπλων και την παρουσίαση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βεβαίω μιας πρότασης οδηγίας για τις κατηγορίες των όπλων. Θα υπάρξει πρόσκληση και προς τη Frontex και τη Europol για εντατικοποίηση των ελέγχων που στόχο θα έχουν την ανείχνευση όπλων και εμπορίου όπλων. Για δε εξωτερικούς ελόγχους στα σύνορα θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν και να υλοποιηθούν συστηματικοί και συντονισμένοι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα. Τους χρειαζόμαστε, το ξέρουμε αυτό. Χρειάζεται να βελτιωθεί μια σειρά μηχανισμών που ήδη υπάρχουν και σε σχέση με την υλοποίηση συστημάτων στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής. Καταχώρηση δηλαδή. Ε, ε, καταγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων κτλ. Θέλουμε να υπάρχει ένα σύστημα αποτελεσματικό, ένα σύστημα με ένα δίκτυο πληροφοριών που θα επιτρέπει την διάγνωση κάθε κίνδυνου και τρομοκρατικής απειλής. Βεβαίως, και αυτό σε σχέση με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου υπάρχουν και στοιχεία για την υιοθέτηση ενός νέου συστήματος, συστήματος Smart Borders όπως ονομάζεται, να τεθεί σε συντονισμό, σε λειτουργία. Πρέπει να μιλήσουμε και για τα smart borders και τη γνωρίζω ότι υπάρχουν ε, ζητήματα και επιφυλάξει από πλευρά τη Επιτροπή σα. Υπάρχουν προτάσεις από πλευρά της Γαλλίας, ιδίως για την ε, αμοιβαιοποίηση των ελέγχων στα σύνορα. Είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως δεν θα συζητηθεί ε, αύριο, Παρασκευή, αλλά στο μέλλον θα πρέπει να το δούμε και να το συστήσουμε εις βάθος. Έκκληση απευθύνεται επίσης στην Frontex στο πλαίσιο των αποστολών της, που είναι κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο της μεταναστευτική πολιτικής, αλλά και στο πλαίσιο αυτό να μην παραγνωρίζει τις πτυχές της καταπολέμησης της τρομοκρατίας κατά τη δράση της. Για την ανταλλαγή πληροφοριών νομίζω ότι ο διευθυντής της Europol είναι ο καταλληλότερος για να σας ενημερώσει. Όπως και η Επιτροπή έχει συμμετάσχει στη διατύπωση των, ε, του σχεδίου συμπερασμάτων που θα υποβάλουμε στο Συμβούλιο για επεξεργασία πρώτα στο Κορεπέρ και μετά στο Συμβούλιο της Προσεχής ώρες. Για τη χρηματοδότηση τρομοκρατίας επίσης, και πάνω απ' όλα τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ, το έχω στα αγγλικά, των Financial Intelligence Units, των ε, υπηρεσιών οικονομικής πληροφόρησης, ε, αλλά και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, απάντηση που θα πρέπει να δοθεί σε επίπεδο ποινική δικαιοσύνης στην τρομοκρατία και τους βίαιους εξτρεμισμούς, θα πρέπει να συντονιστούν οι δυνατότητες που έχουμε και να μετατρέψουμε σε ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και ούτω καθεξής. Και κατά τα άλλα απευθύνουμε έκκληση για δυνατότητες σε προσωπικό, έστω να μπορέσουμε να επιταχύνουμε, να ενισχύσουμε την ανταπόκρισή μας στην, δεν ξέρω μπορώ να πω ακόμα, ή ποια τρομοκρατική επιλή, στον, στην τρομοκρατία που καταρακώνει την Ευρώπη. Αυριανή συνεδρίαση λοιπόν, σύντομα προβλέπεται, λειτουργικού καθαρά χαρακτήρα όπως σας είπα, αλλά βέβαια αληθεύει ότι σε μεταγενέστερο τακτικό συμβούλιο, Τζάι, 4-5 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα, θα επανέλθουμε. Με στοιχεία γενικής πολιτικής, κατά πάσα πιθανότητα, και πιο στρατηγικού χαρακτήρα Ανατολισμός, δεδομένου ότι Τώρα βρισκόμαστε να μια ε, έκτακτη κατάσταση και αυτή και ολούμεθα να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ κύριο Σρούτο. Πρόεδρο, κύριε Κίνα αξιότιμοι βουλευτές, οι αποτρόπες επιθέσεις στο Παρίσι προκάλεσαν γενικευμένο σοκ. Αν δείτε όμως το 2015 είχαμε μια σειρά από επιθέσεις. επτό Κοπενχάγη, το Ταλής και μετά Παρίσι. Διάφορες δημοκρατικές επιθέσεις εκτός Ένωσης και στο Συμβούλιο Τζάι θα υπενθυμίσουν ότι έχουμε και ένα θεματολόγιο για την πολιτική ασφάλεια. Το έχουμε συζητήσει εξάλλου αυτό το ζήτημα επανειλημμένα και εδώ στην Επιτροπή και τα, τους τελευταίους μήνες επικεντρωνόμαστε μάλλον στην ε, μεταναστευτική κρίση και την προσφυγική πρόκληση όπως τον ονομάζω εγώ. Ταυτόχρονα επεξεργαζόμαστε διάφορα στοιχεία του θεματολογίου για την ασφάλεια. Μου ε, έχω διάφορες σημειώσεις εδώ και λένε ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο για διάφορα ζητήματα. Όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσγειωμένοι ε, αν δούμε τι έχει συμβεί ε, στην πραγματικότητα. Με τη Europol ε, έχουμε ε, βελτιώσει τη λειτουργία του δικτύου στο ίντερνετ. Επίσης το δίκτυο της παστικοποίησης είναι μια πρόοδος που έχουμε σημειώσει. Μια νομική βάση για τη ΣΕΠΟΛ που εγκρίναμε πρόσφατα το ώστε να είναι καλύτερη κατάρτιση των ε, αστυνομικών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία αναθεωρημένη ε, εκδοχή του εγχειριδίου Σέγγεν και με τη Europol και άλλους οργανισμούς μπορέσαμε να εντοπίσουμε δείκτες κινδύνου για να βελτιώσουμε τους ελέγχους στα σύνορα. Δεν φτάνει όμως αυτό. Αυτό που προκύπτει από τα γεγονότα. Από την Παρασκευή το βράδυ, Σάββατο το πρωί, ε, έχει ενεργοποιηθεί ο πυρήνας διαχείρισης ε, κρίσεων ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Μπράουν ε, συναντήθηκε με τις Αρχές, τον κύριο Αβραμόπουλο και τον Υπουργό Κασνεύ... για να συζητήσουν την κατάσταση και τώρα έχουμε την αυριανή συνεδρίαση που ακολουθεί. Έχει επιταχύνει τις εργασίες της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εχθές για τα όπλα Το Σώμα των Επιτρόπων υιοθέτησε δέσμη μέτρων για τον έλεγχο κυκλοφορίας των όπλων, ε, καλύπτοντας σε δύο ε, κομμάτια νομοθεσίας. Ένα, ε, θεώρηση της οδηγίας για την αγορά και διάθεση των όπλων, πρέπει να προσαρμόσουμε αυτή τη νομοθεσία και δεύτερον κανονισμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τα κοινά ε, πρότυπα απενεργοποίησης. Χρειαστήκαμε χρόνο για να το καταφέρουμε και χθε ε, συγκαλέσαμε συνεδρίες με του των κρατών για να έχουμε την απαιτούμενη πλειοψηφία και το καταφέραμε αυτό ε, χθε. Ε, κάποια πρόοδο έχουμε κάνει και για τις νομοθετικές προτάσεις. Ε, για το PNR είδαμε το αποτελέσμα του τριμερούς διαλόγου ε, και αυτό με ικανοποίησε, το ανέφερε και ο Κρίστιαν. Πρέπει να δούμε λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα του 11 Φεβρουαρίου του 2015 ότι ελπίζει να ολοκληρωθεί σύντομα ο τριμερής διάλογος και ελπίζω έχουμε έναν λειτουργικό κανονισμό για τη Europol μέχρι το τέλος του 2015. Ε, με παρόδο έχουμε και τη μεταρρύθμιση της ε, προστασίας των προσωπικών δομένων, δεν είναι όμως δική μου αρμοδιότητα και εντάσσεται αυτό στο συνολικό πλαίσιο του επιπρόσθετου ε, πρωτοκόλλου για την Συμβουλία της Ευρώπης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Επίσης, επιταχύνουμε τις εργασίες για την εκπόνηση οδηγίας για την τρομοκρατία ειδικότερα, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εξετάσουμε την απόφαση πλαίσιο που ισχύει τώρα για τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Θα πρέπει τι να υποσχόμαστε να αποφασίσουμε να διοχετεύσουμε και κονδύλια για το κέντρο παραδείγματο χάρη διαχείρισης ε, ε, των κρίσεων και των δημοκρατικών επιθέσεων, υπάρχει αλλά δεν έχει μέσα για να λειτουργήσει. Το κέντρο αντιτρομοκρατία, λοιπόν χρειάζεται κονδύλια και ανταλλαγή πληροφοριών επίση βλέπουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Τώρα, για τα σύνορα, ο πρόεδρος Γιούνκερ είπε ήδη ότι θα καταθέσει πρόταση για τους Ευρωπαίους συνοριοφύλακες μέχρι το τέλος του 2015 να εξετάσουμε το αντίκτυπο επίσης των τρομοκρατικών επιθέσεων για να δούμε αν η έλεγχη για βάση του συνοριακού κώδικα ε, Σέγγεν διεξάγονται όπως πρέπει ή αν χρειάζονται προσαρμογές και το αργότερο μέχρι το Μάρτι του 2016 θα καταθέσουμε πρόταση για τα ευφυή e e σύνορα και τα σημεία εισόδου-εξόδου. Θα δούμε αν θα διατηρηθεί αυτό το φανδιάγραμμα, αλλά προς το παρόν προβλέπεται το αργότερο το Μάρτι του 16. Και πολλά άλλα έχω να σας πω. Νομίζω όμως ότι το ίδιο θα πρέπει επιδιώξουμε πρόοδο για τα περιουσιακά στοιχεία των τρομοκρατικών οργανώσεων. Αύριο στο Συμβούλιο Υπουργών θα συζητηθεί αυτό το ζήτημα. Και πάντοτε είμαι στη διάθεσή σας για να συζητούμε ε, εντελεχέστερα τις προτάσεις. Πολύ σας ευχαριστούμε κύριε Ρούτε. Ε, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ που με προσκαλέσαμε. Είμαστε σαφείς για τις συνέπειες των επιθέσεων της Παρασκευής στο Παρίσι. Εγώ διαπιστώνω μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση των απειλών που έχουμε στην Ευρώπη. Πρόκειται για το πρώτο παράδειγμα στην Ευρώπη επιθέσεως τύπου Μουμπάι με αδιάκριτους πυροβολισμούς εις βάρος πολιτών στο δρόμο και επιθέσεις αυτοκτονίας με βομβιστές, αυτό που φοβόμασταν από το 2008 και το Μουμπάι. Η πραγματικότητα των όσων συνέβησαν στο Μουμπάι τότε ήρθε τώρα πια στην Ευρώπη. Ε, οργανώνεται από ένα ε, διεθνές ε, δίκτυο δραστών που οργανώνονται σε πολλές χώρες και έτσι ορίζεται διαφορετικά πλέον η φύση της τρομοκρατικής απειλής και έχουμε και μια σαφή δήλωση προθέσεων από την ΙΚΙΛ ε, να εξαγάγει τις βίες αυτές επιθέσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κατάρρευση του ρωσικού αεροσκάφους και τις, επιθέσεις, και τις απειλές κατά των ΗΠΑ και άλλες επιθέσεις που γίνονται στην περιοχή γύρω από τη Συρία. Εδώ όμως δεν έχουμε μόνο μια δήλωση προθέσεων, γιατί ξέρουμε ότι έχει σοβαρό δυναμικό και σε ανθρώπινο δυναμικό η ομάδα αυτή και σε υψηλή ε, ποιότητα επικοινωνίας και καινοτομίας χρήση διαδικτύου και κοινωνικών πλατφορμών από την ομάδα. Έχουμε να κάνουμε μια σοβαρή ε, διεθνή τρομοκρατική οργάνωση με πολύ καλούς σπόρους και δικτύωση που είναι δραστήρια τώρα στους δρόμους της Ευρώπης. Και έτσι, χωρίς να θέλω να υπερβάλλω, έχουμε πιθανολόγηση πως μπορούν να συμβούν και άλλες επιθέσεις και είναι η σοβαρότερη απειλή αυτή που αντιμετωπίζει η Ευρώπη τα τελευταία δέκα χρόνια. Από την Παρασκευή το βράδυ κινητοποιήθηκε σε 24 ώρη βάση ε, η υπηρεσία της Europol με διασταύρωση μεγάλου αριθμού δεδομένων που μας ε, χορήγησαν οι αστυνομικές αρχές της Γαλλίας κατά τις ερευνές τους και που αντιπαραβάλλουμε με τη βάση δεδομένων της Europol. Δραστηριοποιούμε την ε, μονάδα ε, παρακολούθησης και διάκρισης στο διαδίκτυο για να εντοπιστούν όχι μόνο πιθανοί δράστες ή υποπτή δράστες, αλλά και πιθανοί μάρτυρες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις γαλλικές αρχές. Πληροφορίες επίσης για τις χρηματικές ροές με το πρόγραμμα TFTP που μας δίνει πάνω από 500 συγκεκριμένε ε, υποδείξεις για διερεύνηση προς τις γαλλικές αρχές αυτή τη στιγμή. Τα πυροβόλα όπλα επίσης που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή την παράνομη αγορά, τη λαθρέα προμήθεια δηλαδή και την πορεία ε, πυροβόλων όπλων προς την Ευρώπη. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι ο κόσμος των εγκληματιών έχει δεσμούς και με την τρομοκρατία Προσπαθούμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό. Έχουμε 625 ενεργές έρευνες αυτή τη στιγμή κατά των εγκληματιών που μπορεί να έχουν κάποια διασύνδεση με την τρομοκρατία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και οι 625 έχουν αποδεδειγμένους δεσμούς, αλλά πάντως έχουμε μια πιο εντατική ε, ε, δραστηριότητα από πλευράς της Europol στο πεδίο της Europol για να διαγνώσουμε αυτές τις απαφές και προσφέρουμε βέβαια και πλατφόρμα αστυνομική συνεργασία σε όλη την Ευρώπη, υποστηρίζοντας και τις γαλλικές έρευνες βεβαίως, αλλά και μια ευρύτερη έρευνα για να δώσουμε μια σαφή ευρωπαϊκή διάσταση στην αντιμετώπιση των επιθέσεων. Έχουμε αποσπασμένους ε, υπαλλήλους στο κέντρο συντονισμού στο Παρίσι τώρα και στις Βρυξέλλες και βέβαια αντίστροφα στα γραφεία της Europol. Έχουμε εντοπίσει μια σειρά από πιθανά ε, πιθανές, ε, ε, εντοπισμού στόχων και πιθανολόγησης που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω διερεύνηση, διασύνδεση μεταξύ τρομοκρατίας και λοιπόν μορφών εγκλήματος, γιατί είδαμε και από τα μέσα ότι καταγράφεται ότι μπορεί να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των τρομοκρατών και ε, κλαπέντο συριακού διαβατηρίου. Οπότε μπορεί να υπάρχουν δεσμοί και με τη μεταναστευτική κρίση και με τα δίκτυα των λαθροδιακινητών. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα ότι υπάρχουν αυτοί οι δεσμοί, αλλά προτεραιότητα της Europol είναι να μελετήσει παραπάνω και να δώσει απαντήσεις. Η σοβαρή βέβαια κλιμάκωση τη απο... της απειλής, είπε και ο πρέσβης ε, Μπράουν, σημαίνουν ότι σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να βελτιστοποιηθεί η αστυνομική συνεργασία και αυτό είναι ο στόχο και του αυριανού συμβουλίου αλλά και στις σημερινές συζήτηση. Η Europol είναι διατεθειμένη να δραματίσει όπω πάντα βέβαια το ρόλο τη, ε, με απόλυτη πληρότητα και επάρκεια. Θα κοιτάξουμε να δούμε πώ μπορούμε να ενισχύσουμε τι εργασίε μα ώστε να δώσουμε καλύτερε υπηρεσίε στι αρμόδιες αρχέ σε όλη την Ευρώπη. Αναβαθμίζουμε ήδη το δυναμικό μα, όπω πει ο κύριο Ρόιτε ε, έχει ήδη ληφθεί απόφαση του Συμβουλίου από την πρώτη στιγμή των επιθέσεων και εμείς ακολουθώντας ε, οργανώνουμε από τις ε, πρώτες μέρες του 2016 ένα κέντρο αντιτρομοκρατικό με συνένωση πορών και βελτίωση του δυναμικού μας σε σχέση με την παρακολούθηση της πορείας της χρηματοδότησης, των εξοπλισμών και βέβαια παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των αλλοδαπών μαχητών για να καταπολεμήσουμε τα δίκτυα της τρομοκρατίας. Προσπαθούμε επίση επίσης να ε, ορίσουμε και ένα συγκεκριμένο αλλά και πολύ διακριτό και διακριτικό πεδίο δράσης και μονάδα που θα ασχολείται μόνο με τη αντιτρομοκρατική δράση. Όπως είπε και ο πρέσβης Μπράουν πρέπει να μεγιστοποιηθεί ιδιαίτερο στο δυναμικό σε ευρωπαϊκή στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανταλλαγή, αποτελεσματική ανταλλαγή των πληροφοριών με στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Έχουμε μεγάλο αριθμό υπόπτων και πολλές χώρες. Είναι πολύ περιπλοκή κατάσταση λοιπόν και έχουμε να κάνουμε με δράστες που πολλές φορές κινούνται μεταξύ τρομοκρατίας και, και σοβαρών εγκληματικών δραστηριοτήτων. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ διαφόρων ε, ειδών και επιπέδων αρχών ώστε να προλαμβάνουμε ε, η αδίποτε σχεδιαζόμενη τροποκρατική επίθεση. Αύριο θα εξετάσει το Συμβούλου αρκετά καταπήγοντα μέτρα και για το PNR, την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων και για τη βελτιστοποίηση του συστήματος ανταλλαγής Schengen και των συστημάτων αντιτρομοκρατικής δράσης και λοιπόν βάσει των δεδομένων της Europol. Εδώ κύριε κλειδί είναι η διαλειτουργικότητα, η διασύνδεση των υπηρεσιών και των πληροφοριών. Βεβαίω θέλουμε ένα πλαίσιο για πιο αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών καθώς είναι πολλαπλές οι βάσει δεδομένων που διαθέτουμε και άρα οι προδιαγραφές για την ασφάλεια πρέπει και να διαφυλιχθούν και να ενισχυθούν με τις υψηλότερου επίπεδου προδιαγραφές ασφαλείας Έχουμε να κάνουμε ένα περίπλοκο έργο, έχουμε να κάνουμε με την ανάγκη για διασύνδεση κατά τρόπο αποτελεσματικό όσο και αναλογικό πολλαπλών βάσεων και επιπέδων για να έχουμε στο δυνατόν ασφαλή αλλά και βέλτιστη ε, λειτουργία. Στον χώρο των αντιτρομοκρατικών, η Europol προς τα τελευταία χρόνια προσπαθούσε πάντα να κινητοποιήσει τις εθνικές αρχές να διαθέτουν τις πληροφορίες τους σχετικές με τρομοκρατικές απειλές μέσω της Europol στους, στους λοιπούς εταίρους και όχι μόνο για τις πιο προβεβλημένες έρευνες όπως πράττει τώρα η Γαλλία αλλά και με τρόπο συστηματικό που θα λειτουργήσει προληπτικά. Έχουμε σημειώσει σημαντικές βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια αλλά όπως είπε ο κύριος Ρούτ δεν έχουμε ε, ολοκληρώσει αυτό το έργο και ιδιαίτερα Έχουμε μία βάση δεδομένων για τους ταξιδιώτες ε, που καταγράφει τις κινήσεις υπόπτων ε, αλλοδαπών μαχητών ε, από τη Συρία και το Ιράκ μέσα στην Ευρώπη. Με 10.000 περίπου υπόπτους, εισόδους καταγεγραμμένες από τα κράτη-μέλη και τους διεθνείς εταίρους. Τελευταίους δύο μήνες έχουν διπλασιαστεί τα νούμερα αυτά. Αυτό είναι ήδη θετικό μήνυμα. Βέβαια οι 2.000 από τις 10 αυτές μπορούν να, μπορεί να βεβαιωθεί ότι είναι, ότι είναι όντως αλλοδαποί μαχητές, οι υπόλοιποι όμως είτε έχουν εμπλακεί στη διευκόλυνση της διακίνησης αυτών των αλλοδαπών μαχητών είτε μπορεί να είναι ύποπτοι ε, μαχητές. Άρα λοιπόν χρειάζεται περαιτέρω μελέτη. Πάντως υπάρχουν 5.000 Ευρωπαίοι υπήκοοι που ταξιδεύουν ε, στο Ιράκ και τη Συρία αυτή τη στιγμή. Όλες οι είσοδοι περνούν από 5 κράτη-μέλη και έναν άλλο διεθνή εταίρο. Άρα χρειάζεται αυτή η επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών. Τώρα που υπάρχει ε, η που είναι η κατάλληλη στιγμή πρέπει να κινητοποιήσουμε όλες τις αρμόδιες αρχές πρέπει να δώσουμε νέες δυνατότητες για διαλειτουργικές πλατφόρμες τις οποίες θα μπορούν οι αρμόδιοι για την αντιτρομοκρατική δράση, αξιωματούχοι από διάφορε υπηρεσίες να συμμετέχουν, να προσφέρουν πληροφορίες, να δίνουν ε, τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη για απόσπαση προσωπικού σε αυτή την πλατφόρμα. Αύριο θα συζητήσουμε την πιο συστηματική χρήση του συστήματος πληροφοριών Schengen για να ε, εξασφαλίσουμε και την βέλτιστη δηλαδή στελέχωση από πλευρά των κρατών μελών και βέβαια σε συσχετισμό μεταξύ του συστήματος πληροφοριών Schengen και της βάσης δεδομένων της Europol. Στα εξωτερικά επίσης σύνορα με, την περιφερειακή, με τις περιφερειακές task force στην Ελλάδα και την Ιταλία ε, αλλά και σε ευρύτερη συνεργασία με τα κράτη-μέλη για μια πιο αποτελεσματική ε, καταχώρηση και εξέταση των υποψηφίων ε, για ε, διάβαση των συνόρων. Θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Δίεστε Μέρα για την δραστήρια συμμετοχή του στον τριμερή διάλογο. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τα λόγια του. Είναι κατεπίγουσα η ανάγκη να ολοκληρωθούν οι προτάσεις αυτές το χειτερό δυνατό. Πρέπει βεβαίως να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο και συνέπεια θα εξασφαλίσει σε σχέση με τις ανάγκες ε, της Europol να στηρίξει την αντιτρομοκρατική δράση των κρατών μελών, να προστατεύσει τους πολίτες από την απειλή της ε, τρομοκρατίας στο χέτερο δυνατό και ιδιαίτερα θέλω να υπογραμμίσω την ανάγκη για μια αποτελεσματική βάση δεδομένων το χέτερο δυνατό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Thank you for all Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Συνάδελφοι, ξεκινάμε την συζήτηση. Πολλοί από σας ζητήσατε το λόγο, θα σας ε, το δώσω και μετά. Θα κλείσουμε το κατάλογο. Έχουμε τους συντονιστές, Χολμάιερ. And Mrs. Meyer. And then Στη συνέχεια, Mrs. Revaud-Dallon, Mrs. Guillaume, Mrs. Gomez, Mrs. Vergia, Mrs. Lauristin, Mrs. Wimberg, Mr. Albrecht, Mr. Mello, Mr. Weidenholzer, Mr. Jurek, and that's all. Now I close the list. I will ask all you, all of you, to keep to a two minutes time frame, time limit. Otherwise... Λοιπόν, θα έχουμε δύο λεπτά χρόνο, χρόνο έκαστος, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις τον προσκεκλημένο μας. Πρώτα οι συντονιστές, η κυρία Χολμάγερ. ζητώ συγγνώμη γιατί δεν θα μπορέσω και το λέω προκαταβολικά να τήρξω το χρόνο γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία το θέμα αυτό και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα ήθελα να εκφράσω ότι βαθύτατα συλληπιτήριά μου προ τι οικογένειε πάνω απ' όλα και του οικείου των θυμάτων. Είναι απαραίτητο αυτό να το πράξουμε σε τέτοια χρονική στιγμή. Και ιδιαίτερα θέλω να εκφράσω τι ευχαριστίε μου και το μέγιστο σεβασμό μου στι αρχέ ασφαλεία τη Γαλλία, ιδιαίτερα για το πολύ δύσκολο έργο το οποίο επιτελούν, επικίνδυνο και δύσκολο έργο που επιτελούν τι τελευταίε ημέρε. Και ίσω θα έπρεπε ω Επιτροπή Πρόεδρε, μέσω ημών να αποστείλουμε μια επιστολή στον Υπουργό Κασνεύ για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη και την αναγνώρισή μας για αυτές τις προσπάθειες. Νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε σε αυτή τη χρονιστική στιγμή ότι είναι πολύ ότι ε, αναγνωρίζουμε και δείχνουμε ευγνωμοσύνη για αυτή τη δράση. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα. Θα ήθελα, ε, αγαπητέ κύριε Πρέσβη, να ρωτήσω για το Συμβούλιο. Είπατε ότι θα γίνει την Παρασκευή αυτή η συνεδρία. Θα ήταν πολύ καλό και η Επιτροπή μαζί με σας να μας ενημερώσει αμέσως μετά, Δευτέρα δηλαδή, ή αν όχι, την παραπάνω εβδομάδα για να γνωρίζουμε τι αποφάσεις έχουν ληφθεί έτσι ώστε και η δική μας η Επιτροπή να ε, προχωρήσει μια ταχύτατη και συντονισμένη συνεργασία για να υποστηρίξουμε ενδεχόμενα μέτρα που θα χρειαστεί να συζητηθούν. Πολλά είναι τα μέτρα τα οποία ε, μας έχουν ήδη απασχολήσει εδώ και αρκετό χρόνο, άρα δεν είμαστε σε μια βεβαιασμένη δράση. Δεν είναι κάτι το καινούριο το θέμα και η συζήτηση για την προστασία των συνόρων, ε, δεν είναι κάτι το καινοφανές, αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε την ενημέρωση για να μπορέσουμε στοχευμένα να συζητήσουμε και να συνεργαστούμε. Πάλι με το σύστημα PNR για την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων βρισκόμαστε σε ένα γνωστό πεδίο Πρέπει όμως να προχωρήσουμε και γι' αυτό θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι ε, θέσεις έχει διατυπώσει το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Τι προγραμματίζεται για δράση. Για να αναφερθώ στα λόγια του κυρίου Ρέιτς. Και πάλι επισημαίνεται το πρόβλημα της επάνδρωσης της Europol για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας όπως και για την καταπολέμηση των πιο σοβαρών μορφών εγκλημάτων. και σε αυτό ως Επιτροπή και εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος το διατυπώνω επίσημα ως πρόταση κυρία Πρόεδρε, θέλουμε μια φορά το χρόνο να μας αποδίδεται μια έκθεση για την κατάσταση ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορούμε τακτικά με τη μορφή αυτών των ακροάσεων να ενημερωνόμαστε και να διατυπώνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Μέσα σε ένα τέταρτο που ε, μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας για να ενημερωθούμε για τα όσα συμβαίνουν στα κράτη-μέλη. Προφανώς δεν μπορούμε να πούμε και να μάθουμε αρκετά. Και ο κύριος ε, Δίες Δεμέρα και άλλοι συνάδελφοι έχουν ε, ζητήσει να ενημερωνόμαστε από τη Europol αλλά και από τις υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών μελών τακτικά εδώ στην Επιτροπή μας, ώστε να έχουμε κάτι συγκεκριμένο ως Επιτροπή κάτι συγκεκριμένο για την συγκεκριμένη κατάσταση όπως υπάρχει, γιατί είμαστε σε μεγάλη απόσταση, ζούμε σε μεγάλη απόσταση από την πραγματικότητα και χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες σχετικές με την πραγματικότητα και να βρεθεί ασφαλώς ο χρόνος από τις συνεδριάσεις μας για την ουσιαστική συζήτηση. Όχι, όχι μια ώρα μόνο, ε, στοχευμένα να μπορούμε να δούμε διαφορετικούς τομείς ε, για τους οποίους θα μας δοθούν συγκεκριμένες πληροφορίες, να διαγνώσουμε πού υπάρχουν κενά ασφάλειας, τι έχει εντοπιστεί, τι γνώσεις έχετε, γιατί συμφωνώ απολύτως ε, σε αυτά που είπατε βεβαίως, αλλά ίσως αν είχαμε και περισσότερες πληροφορίες θα μπορούσαμε ως Επιτροπή να λαμβάνουμε πιο αποτελεσματικά και στοχευμένα τις αποφάσεις μας για την ομοθεσία. Και κάτι ακόμη το οποίο με προβληματίζει ιδιαίτερος και πάλι μας λείπουν πληροφορίες και ενημέρωση. Θέλω να ρωτήσω σε ποιο βαθμό μπορούν οι τρομοκράτες να αξιοποιήσουν συστήματα κωδικοποίησης ώστε ακόμη και κατά τη διάρκεια των τρομοκρατικών επιθέσεων να μπορούν να ξεφεύγουν από την επιτήρηση των αστυνομικών αρχών. Είναι πολλά τα ερωτήματα που έχω. Λοιπόν, συμφωνώ με το PNR, για την οδηγία PNR και για την οδηγία Europol και για τα ζητήματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων πρέπει να εξοργανωθεί το ταχύτερο δυνατό μία συζήτηση. Είτε για τους κανονισμούς είτε για τις οδηγίες πρέπει να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό ε, χωρίς αντιπαραθέσεις, με μια ουσιαστική διαδικασία συζητήσεως διαρθρωμένη, στην οποία θα συμμετάσχουμε όλοι και θα προωθήσουμε το ταχύτερο δυνατό τα ζητήματα αυτά. Ε, παρακαλώ λοιπόν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ξέρω ότι η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να επιταχύνει πολλού ρυθμού τη, αλλά το ταχύτερο δυνατό πρέπει να δράσει. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μπράουν και ο κύριο Ρούτε πρέπει να πάνε στην Κορεπέρ. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακούσουμε του συντονιστέ και μετά από το γύρο των συντονιστών θα του καλέσουμε να απαντήσουν. Οι υπόλοιπε παρεμβάσει των συναδέλφων θα ακολουθήσουν. Η κυρία Ένστε. Nein, äh, für unsere Fraktion spricht Frau... Äh, Όχι, εκ μέρου τη ομάδα μα θα λάβει το λόγο η κυρία Βεργιά. Εγώ είχα ζητήσει το λόγο ω λυπή ομιλήτρια. Έτσι αποφασίσαμε. Merci, Madame la... Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω σας ευχαριστώντας σε όλους για την αλληλεγγύη που επιδείξατε. Νομίζω πως ακόμα η συγκίνηση επικρατεί, αλλά θα ήθελα, όπως είπε και η κυρία Χολμάγερ, να σκεφτούμε πρώτα ναι, τα θύματα και τις οικογένειές τους και να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν στη διάρκεια της Παρασκευής και της νύχτας της Παρασκευής προς το Σάββατο, αστυνομική, πυροσβεστική και ε, προσωπικό υγιές που όλη τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού έκανε εξαιρετικό έργο, έσωσε ζωές και εξακολουθεί να το κάνει. Πιστεύω πως είναι φυσιολογικό μια κυβέρνηση να αντιδράσει απέναντι στη φρίκη των όσων ε, συνέβησαν την Παρασκευή που έπληξαν καταρχήν νέους, νέους διαφόρων εθνικότητων, πολλούς Γάλλους βέβαια, αλλά και άλλους Ευρωπαίους και όχι μόνο Ευρωπαίους. Και καλό είναι αυτό να το θυμίσουμε. Ε, το, το, η Νταέσ ήδη είχε χτυπήσει το Παρίσι και υπήρξε και, υπήρξαν και οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Πυρητόλα και το ρωσικό αεροπλάνο στην Αίγυπτο. Υπήρξαν, ε, ε, αυτές οι επιθέσεις ε, στα τυφλά έγιναν, στόχευσαν στα τυφλά. Αυτό έχει ξανασυμβεί παλιότερα, γιατί εφόσον έχω μια κάποια ηλικία, θα θυμίσω ότι υπήρξαν τρομοκρατικές επιθέσεις στη δεκαετία του 80, του 90, στο Παρίσι αλλά και στη Μαδίτη και στο, Λονδίνο. Και εκεί τυφλές ήταν οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Πολλοί κόσμοι σήμερα φοβάται, φυσικό είναι. Και βέβαια ε, θα πρέπει να φροντίσουμε για την ασφάλεια όλων και καθενό χωριστά. Και ξέρουμε όλοι ότι ο μηδενικό κίνδυνο δεν υπάρχει. Ναι, πρέπει να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, ναι, να καθησυχάσουμε τον πληθυσμό, ναι, να τον προστατέψουμε. Αλλά εμένα με εντυπωσίασε η ατμόσφαιρα που επικρατεί στη Γαλλία και κυρίως στην ε, διαφορά ανάμεσα στο κλίμα που επικράτησε μετά το Σαρλί και μετά το... Και, τώρα. Πολλοί κόσμος λέει θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε φυσιολογικά, διότι δείχνοντας ε, ότι φοβόμαστε και ότι έχουμε πανικοκληθεί, παίζουμε το παιχνίδι του Νταές. Και πιστεύω πως αυτό, αυτή η σκέψη, το είδαμε και αυτό το βράδυ, στη Μόλεμπεκ, είναι μια υγιής αντίδραση σε μια δημοκρατία και σε ένα κράτος δικαίου. Πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε την επιζυχρεμία μας και τη λογική μας και να θυμίσουμε τις βασικές μας αρχές που ανέκαθεν ε, μας καθοδήγησαν εδώ σε αυτή την Επιτροπή και κυρίως ε, η αρχή της ε, αναλογικότητας και της ανάγκης από τη στιγμή που θίγονται και θεμελιώδεις ε, ελευθερίες. Και έχω να κάνει κάποιες παρατηρήσεις, θα πάω γρήγορα. Βέβαια πρέπει να συγχαίουμε τα επίγοντα μέτρα με τα πιο μακροπρόθεσμα. Να υπογραμμίσουμε ότι στα όσα είδαμε την Παρασκευή περισσότεροι εγκληματίε αυτοί είναι Γάλλοι υπήκοοι και όπως και τον Ιανουάριο αυτό το οποίο προτάσσεται είναι το θέμα του συντονισμού σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Δεν ξεχνώ ότι τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο ένας από αυτούς τους τρομοκράτες διέσχισε τα γαλλοβελγικά σύνορα και μάλιστα τον σταμάτησαν οι αστυνομικέ δυνάμεις χωρίς να τον συλλάβουν να ε, ανησυχώ για την εφαρμογή του PNR και του Smart Border που μας παρουσιάστηκε αρχικά ως ένα εργαλείο για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των τουριστών, έπειτα ως ένα εργαλείο κατά της μετανάστευσης και τώρα κατά της τρομοκρατίας. Εγώ πιστεύω πως όλα αυτά τα μέσα κοστίζουν ε, κολοσσία ποσά και ότι το κεντρικό πρόβλημα που υπάρχει είναι η ανάγκη για ανθρώπινους πόρους. Αυτό απεδείχθη δυστυχώς και στο Παρίσι ε, και ανησυχώ επίσης για το συστηματική σύνδεση που γίνεται ανάμεσα στην καταπολέμηση του τρομοκρατίας και την μετανάστευση. Οι πρόσφυγες στη Σύρη είναι το πρώτο και κύριο θύμα του Νταές. πρέπει να το θυμίσω αυτό και να κάνω και μια παράθεση του Βενιαμίνου Φραγκλίνου ότι ένας λαός ε, που θυσιάζει την ελευθερία του για μεγαλύτερη ασφάλεια δεν αξίζει το ένα το άλλο και θα καταλήξει χάνοντας και τα δύο. Αυτή τη φράση πρέπει να την έχουμε διαρκώς στο μυαλό μας και να μας καθοδηγεί ώστε να ε, ε, κρατήσουμε λογική, τη λογική μας μετά από όλα αυτά γιατί διαφορετικά θα παίξουμε το παιχνίδι του Νταές. Η κυρία Λαουριστίν μου είπαν ότι θέλει να μιλήσει εξ των σοσιαλιστών, σοσιαλδημοκρατών. Θα ήθελα να σας πω ότι θα μιλήσουν οι συντονιστές. Αλλά να ξέρετε ότι τρώτε το χρόνο των συναδέλφων, γιατί κάποια στιγμή τελειώνει αυτή η συνεδρίαση, έχει όριο. Ε, κυρία Λαουριστίν, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό που έχω να πω από, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών είναι ότι η κατάσταση μετά την Παρασκευή έχει αλλάξει πολύ. Ε, στο Έχει αλλάξει και το πλαίσιο της δουλειάς που κάνουμε αμφίδρομα. Από τη μια πλευρά καταλαβαίνουμε ότι σε αυτή την κατάσταση γίνονται συγκεκριμένες προσπάθειες ε, από πλευράς όλων των θεσμών που ασχολούνται με την ασφάλεια και την κατασκοπία ε, τη συλλογή πληροφοριών. Αυτά είναι όλα επίγοντα. Αυτά τα στηρίζουμε φυσικά, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο μια τρομοκρατική επίθεση ε, σαν να είναι κάποιο ε, τρομοκρατική οργάνωση που κυκλοφορεί σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά είναι πολύ σαφείς δραστηριότητες του κράτους, κρατη, μάλλον ενός ε, αυτοοριζόμενου κράτους ε, ίσης, του Ισλαμικού κράτους ή του Νταές, που αυτή τη στιγμή ε, μετατρέπεται στο πιο σημαντικό εχθρό, όχι μόνο για τη Γαλλία. Η Γαλλία είναι συμβολικό το πρώτο μέρος το οποίο δέχεται επιθέσεις, λόγω του ότι σαρκώνει τις ευρωπαϊκές αξίες κατά κάποιο τρόπο, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρόκειται για επίθεση κατά της Ένωσης και των αξιών της και αυτές είναι οι αξίες που πρέπει να προστατεύσουμε καταρχάς και είναι η ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία και ούτω καθεξής. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Βερζιά για την πολύ συγκεκριμένη αντίδραση του κόσμου στη Γαλλία που σαφώς καταλαβαίνει τι διακυβεύεται εδώ. Διακυβεύονται οι ελευθερίες μας, ο τρόπος ζωής μας, οι αξίες μας αυτού του είδους η ασφάλεια που γίνεται μέσω της, ανθρω... της προστασίας της ανθρωπιάς. Και εδώ βεβαίως θα πρέπει να κατανοήσουμε και να διατηρήσουμε την ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και αυτές τις αξίες. Αυτό είναι το βασικό μας καθήκον σε αυτόν τον αγώνα κατά του ΝΤΑΕΣ. συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη είναι το πιο σημαντικό. Η Γαλλία ζήτηση ελληνική και είμαστε έτοιμοι να την προσφέρουμε. Αλλά ποια είναι τα συγκεκριμένα εργαλεία, τα μέσα που έχουμε, αφού ακούσαμε και από τον κύριο Πόλα ότι για παράδειγμα μόνο πέντε χώρε έχουν ε, πάρει σοβαρά ε, υπόψη τι ευθύνε του για να ανταλλάσσουν πληροφορίε. Το πρόβλημα λοιπόν με την ανταλλαγή πληροφοριών και με την ε, παγιωμένη δράση ανάμεσα στα κάτι μέλη οριζόντια είναι το πιο σημαντικό που θα πρέπει να βελτιωθεί. Και σε αυτό το πλαίσιο θέλω να τονίσω ότι ο συγητής ότι η οδηγία είναι ένας τρόπος ώστε να έχουμε περισσότερους ξεκαθαρούς κοινού κανόνες που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την επιβολή του νόμου σε όλα τα κρατημέλη, για να ανταλλάσσονται πληροφορίες, να γίνονται συντονισμένες δράσεις, να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στα κρατημέλη και τη Γεροπόλ και ούτω καθεξής. Θα πρέπει δηλαδή να συνεχίσουμε το πλαίσιο είναι το ίδιο και οι αξίες είναι οι ίδιες. Ευχαριστώ. Thank you. Mrs. Sargentini, please. Η κυρία Σαργεντίνη, παρακαλώ. Ένα από τους ομιλητές είπε ότι οι προτάσεις που έγιναν για τις αποφα... και οι αποφάσεις που ελήφθησαν μετά τι επιθέσει τη Charlie Hebdo δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν μετά από τι επιθέσει τη Charlie Hebdo. Και αυτό είναι Αυτές που και αυτές που στηρίζω είναι λυπηρό αυτό και για τις άλλες όχι. Ε, αλλά κάτι που έπρεπε να κάνουμε μετά από το... Σε επιθέσεις του Τσαρλί Εμπντό, ε, είναι το δίκτυο για την ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή, ε, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενημέρωσης για τις ριζοσπαστικοποίησει. Αποφασίστηκε να δημιουργηθεί αυτό το δίκτυο για να, ε, για να βοηθηθούν άνθρωποι που δουλεύουν στις ε, φυλακές, ε, οι αστυνομικοί, οι εργαζόμενοι με τους νέους, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν και να ενημερώνουν κατά πόσο κάποιος ριζοσπαστικοποιείται και να προσπαθήσει να βρει τα λόγια για να το αντιστρέψει αυτή την κατάσταση, να εργαστεί δηλαδή για να αποτραπεί αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στην Ευρώπη και πριν από λίγους μήνες έμεινε χωρίς χρήματα, γιατί και πάλι είδαμε ότι στο Παρίσι τρομακτικά Ευρωπαίοι υπήκοοι. Μεγάλωσαν εδώ στην Ευρώπη, ε, μορφώθηκαν στην Ευρώπη, ριζοσπαστικοποιήθηκαν στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει και η απορριζοσπαστικοποίηση. για να ε, μπορέσουμε να έχουμε αυτό το δίκτυο ε, και να ε, λειτουργήσει, να κάνει πολύ περισσότερα. Συμφωνώ με τον Διευθυντή της Europol ότι η ανταλλαγή των πληροφοριών ανάμεσα στους οργανισμούς ασφάλειας και της αστυνόμευσης είναι πολύ σημαντική. Εδώ έγινε επίθεση κατά του Μουσείου, Εβραϊκού Μουσείου πέρυσι και διαπιστώσαμε ότι οι γαλλικές υπηρεσίες γνώριζαν τον τύπο αυτό, και, αλλά κανείς δεν ενημέρωσε τους Βέλγους. Τώρα πάλι βλέπουμε ότι οι Βέλγοι ξέραν περισσότερα για αυτούς τους ανθρώπους που επιτέθηκαν στο Παρίσι, αλλά ποτέ δεν είπαν στους Γάλλους. Μα... Λέγεται ότι θέλετε για PNR και για τις μεγάλες βάσεις δεδομένων, αλλά το κύριο είναι ότι υπάρχουν υπηρεσίες ασφάλειας που τις συγκεντρώνουν τις πληροφορίες αλλά δεν τις δίνουν. Αν αυτό δεν λυθεί δεν κάνουμε τίποτα, μια τρύπα στο νερό. Από ριζοσπαστικοποίηση, επιτόπου αστυνόμευση, συλλογή, όχι συλλογή πληροφοριών, ανταλλαγή πληροφοριών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η φιλελεύθερη παρακαλώ. Κυρία Παγασάουρ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι στην Ισπανία θυμόμαστε πολύ καλύτερα το πώς τις τρομοκρατικές επιθέσεις γιατί μια σημαντική πολιτι... πολύ σημαντική πολιτική γλίτωσαν από τρομοκρατικές επιθέσεις ε, και πιστεύω πως θα μπορούσαμε να το αντιληφθούμε με πολύ πολύ έντονο τρόπο το τι γίνεται. Κάτι τόσο οργανωμένο όπως αυτό που συνέβη στο Παρίσι μας ε, κάνει να Ε, λέμε ότι ναι, θέλουμε όλα τα απαραίτητα μέσα, αλλά όταν μιλάμε για τα επίγοντα και τα σημαντικά θα πρέπει να θυμίσουμε από τη μια πλευρά ότι η Europol χρειάζεται όλα τα, μέση, τα μέσα ε, ότι τα κράτη πρέπει να έχουν την πολιτική βούληση να συνεργαστούν πολύ πιο εντατικά από ό,τι μέχρι τώρα και ότι όντως μεσοπρόθεσμα είναι απαραίτητο ε, να γίνει δουλειά προληπτική, πρόληψης. Μόνο το ένας αστυνόμος δεν μπορεί να τα καταφέρει να αντιμετωπίσει ένα κίνημα ένα τεράστιο κύμα φανατισμού. Μόνο αστυνομεύοντας δεν γίνεται. Είναι σημαντικό. Χωρίς πρόληψη δεν πρόκειται να μπορέσουμε να ξεμπερδέψουμε με αυτή την υπόθεση. Και τα δυο λοιπόν είναι σημαντικά, είναι απαραίτητα. Χρειάζονται περισσότερα χρήματα και περισσότερη πολιτική βούληση. Η Europol χρειάζεται δική μας στήριξη. Όλοι, όλοι θέλουν στήριξη. Από πλευράς των φιλελευθέρων θα την έχετε. Θέλω αυτό να το πω ξεκάθαρα, γιατί πρόκειται για μια απειλή τέτοιου επίπεδου που το φοβόμασταν, αλλά που όλα, έφτασε και όλα στην Ευρώπη. Είμαστε όπως στη Βομβάη το 2012. Η κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω, ξεκινώντας εξ ονόματος της ομάδας μου, να εκφράσω την ε, βαθύτατη συντριβή μου για τα θύματα του Παρισιού. Εκ μέρους της Προεδρίας του Συμβουλίου μίλησε ο εκπρόσωπος για την, απόφαση, για την συνεδρίαση που πρόκειται να διεξαχθεί αύριο την Παρασκευή. Θα ήθελα να ρωτήσω τι λέει για, την, για μια πρόταση να απαγορευθεί η πώληση πυροβόλων όπλων, να προτείνει δηλαδή στα κράτη-μέλη ένα εμπάργο στην πώληση πυροβόλων όπλων, μιλήσατε για τη διάγνωση κτλ. Γιατί δεν απαγορεύεται την ε, πώληση των όπλων και όταν μιλούμε για, τον κύριο, για την κύρια πηγή τροφοδοσίας αυτών των πολέμων, γιατί να μην προσπαθήσουμε να τους λύσουμε, να λύσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του, αντί να προσπαθούμε να καλύπτουμε ε, με μπαλώματα, με εμβαλωματικέ λύσεις ε, τα προβλήματα. Δεν πρέπει να βρούμε μια ουσιαστική λύση και σε αυτό να κερδίσουμε τα κράτη-μέλη. Για δε την ανταλλαγή πληροφοριών που ανεγνωρισμένα σήμερα έχει αποτύχει ή πάντως δεν είναι αποτελεσματική. Έχουν εντοπιστεί κοινοί δείκτες κινδύνου. Αλλά πέραν αυτού δεν ε, υπάρχει η αναγνώριση των περαιτέρω δράσεων που θα χρειαστούν. Χωρίς να θέλω λοιπόν να προβώ σε ε, ε, επικριτική αντιπαράθεση, θα θέλω να ρωτήσω γιατί δεν λειτουργήσε αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι ζήτημα επικοινωνίας μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, ε, απουσίας επικοινωνίας, επιφυλακτικότητας ως προς τη διάθεση πληροφοριών ή το σύστημα όπως έχει σχεδιαστεί δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί προφανώς υπάρχει κάποιο κενό, κάποιο έλλειμμα στην ανταλλαγή των πληροφοριών μέσα στο ίδιο το σύστημα. Και δεν μπορούν και να αξιοποιηθούν πληροφορίες που ενδεχομένω λαμβάνονται και να αναλυφθούν δράσεις συγκεκριμένε στη συνέχεια. Για δε την εντατικοποίηση των ελέγχων στα σύνορα και πιθανή διασύνδεση με λαθροδιακινητές ε, και σωματεμπόρους ή εμπόρους ανθρώπων. Λέτε ότι πρέπει να αντείνονται οι έλεγχοι, να πολλαπλασιάζονται οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα και να, ενταθούν, να ενταθεί η παρουσία των αρχών φύλαξη των σύνορων. Αλλά οι ετούντες του άσυλο θα έχουν τη δυνατότητα να φτάνουν στην Ευρώπη με τρόπο νόμιμο και ασφαλή. Γιατί οι λαθροδιακινητές, εάν τους αναφήναμε ένα νόμιμο δρόμο εισόδου για τους πρόσφυγες θα έχαναν την πηγή των εσόδων τους, θα καταπολεμούσαμε έτσι το πρόβλημα στην πηγή του και βεβαίως ταυτόχρονα θα με τον πιθανό σύνδεσμο μεταξύ αυτών των λαθροδιακινητών και της τρομοκρατίας συγκεκριμένα και καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως τον ε, δόκτωρα Ρούιτε να μας πει τι γνώμη έχει γι' αυτό, γιατί δεν βλέπουμε ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς να έχει ε, δώσει πιο συγκεκριμένες προτάσεις, ενώ μιλούσε για το άνοιγμα των θυρών ε, διόδου προς την Ευρώπη. Δεν έχουμε δει πιο συγκεκριμένε προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει η περίπτωση, μελετάτε μια τέτοια αριθμιστική παρέμβαση. Γιατί για το Δουβλίνο γίνεται λόγο, ενώπιση του Δουβλίνου γίνεται λόγος για διαφορετικές λύσεις, μέτρα τα οποία δεν θα εξασφαλίσουν όμως νόμιμη είσοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για τις οικογένειες ε, των θυμάτων πραγματικά εξοργίζομαι με τους θανάτους αθώων εξαιτίας ε, Ισλαμιστών τρομοκρατών. δεν έχουν καμία σχέση με το Ισλάμ, ε, από το Ισλαμικό κράτος. Ε, είναι ε, στρατιώτες ενός παράνομου κράτους, άνεργοι άνθρωποι που βρίσκονται σε απόγνωση, δεν έχουν καμία σχέση με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναρωτιέμαι το εξής, ε, τι κάνετε εσείς, ε, πόσοι ακόμη αθώοι θα πρέπει να πεθάνουν προτού κινηθούμε, ε, κινητοποιηθούμε. Πρόκειται για την ασφάλεια των πολιτών που εμείς εκπροσωπούμε. Μιλάμε για μέτρα, αλλά πρέπει επιτέλους να τα εφαρμόσουμε. Θα ήθελα να κάνω λοιπόν εγώ δύο συγκεκριμένες προτάσεις. Να αποεσλαμικοποιήσουμε τα κράτη-μέλη Επιστρέφω στους προσκεκλισμένους μας για να δώσουμε τις απαντήσεις. Ο πρέσβης Μπράουν και στη συνέχεια ο κύριος Ρούτε. Παρακαλώ. Ο κύριος Μπράουν. Ε, θα απαντήσω τις ε, ερωτήσεις με τη σειρά. Κυρία Χολμάιερ, ε, πάντοτε είμαστε στη διάθεσή σας για ένα debriefing. Ακόμη και αν δεν έρθουν οι υπουργοί, θα έρθω εγώ αυτοπροσώπως. Έχουμε καλέσει τον πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για το γεύμα την Παρασκευή για να γίνει ανταλλαγή απόψεων με τους υπουργούς εσωτερικών. Για το PNR Είπατε ότι δεν κεγόμαστε τώρα γιατί δεν είναι κάτι καινούριο αυτό το ζήτημα. Εγώ θα έλεγα όμως ότι πρέπει να σπεύσουμε και να το, και να το προχωρήσουμε. Υπάρχουν θέματα που συνδέονται όχι άμεσα, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ένα πακέτο. Το Κοινοβούλιο ζήτησε να είναι πακέτο όλα αυτά τα ζητήματα και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Είναι σημαντικό να ε, υποστηρίξουμε όλο αυτό το πακέτο. Νομίζω ότι λόγω της ε, κατάστασης πρέπει να έχουμε κάτι να προσφέρουμε στην, ε, στους πολίτες μας. Να δείξουμε ότι δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά. Για τις ε, επιχειρησιακές ε, διαστάσεις έχουμε ήδη κάνει διάφορες συναντήσεις ε, για το κόζι παραδείγματος χάρη και έχουν γίνει και συναντήσεις στις Βρυξέλλες αυτών που είναι αρμόδιοι για τις υπηρεσίες πληροφοριών. για την ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, φυσικά όλα αυτά γίνονται ε, με μυστικότητα για ευνόητους λόγους, αλλά υπάρχει κινητοποίηση. Κυρία Βεζιά. Σωστά τα λέτε. Ε, πρέπει να προστατεύσουμε το κράτος δικαίου, το οποίο όμως δέχτηκε επίθεση από τους τρομοκράτες με εξαιρετικά ομό βίο και απάνθρωπε τρόπο. Χρειαζόμαστε μια αναλογικότητα στην απόκριση που δίνουμε σε τέτοιες επιθέσεις. Ε, σε σχέση με την κυρία Λαριστίν πρέπει όντως να προσπίσουμε τις αξίες μας σε την αξία της ελευθερίας αλλά θα πρέπει να είναι ασφαλείς οι πολίτες. Πρέπει να βρούμε την ε, ισορροπία ανάμεσα στα δύο και είστε εισηγήτρια για αυτό το ζήτημα. Θα παρακολουθήσετε στενά αυτά που κάνουμε. Η κυρία Σαρτζεντίνη, σπαστικοποίηση, είναι και δύσκολη η λέξη. Θα το συζητήσουμε στην, ε, στο Συμβούλιο Υπουργών την Παρασκευή. Έχουμε καλέσει και τους Υπουργούς Δικαιοσύνης. Ε, Ορτοάντο, ε, κάνατε μάλλον μια πολιτική δήλωση, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας ως επιτοπλίστων. Κυρία Φεράρα, για την ανταλλαγή πληροφοριών, όντως αν έχετε το καλύτερο δυνατό ε, σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, πάντοτε θα υπάρξουν στιγμές που δεν ε, θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα. 5.000 ε, αλλαπούς μαχητές ε, είχαμε και ξέρουμε ότι ήδη έχουμε αποτρέψει πάρα πολλές επιθέσεις χάρη σε αυτές τις πληροφορίες, όμως χρειάζονται μετατικότερες προσπάθειες και αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα για τους υπουργούς το, την Παρασκευή, όχι για την ανταλλαγή πληροφοριών σε σωστό επίπεδο, αλλά για την προώθηση των πληροφοριών και την πίεση ε, προς τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να συνεργαστούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Για τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης, όχι, δεν το ξεχάσαμε. Αυτή την εβδομάδα καταλήγουμε συμφωνία για τους ε, ε, φοιτητές ερευνητές. Δεν προβάλλεται το ζήτημα διότι είναι τραγικές οι συνθήκες που επικρατούν λόγω των περιστατικών, αλλά όλα προχωρούν και θα σας ενημερώνουμε για τους συνοριακούς ελέγχους. Ε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρούτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο. Δεν θα επαναλάβω όλες τις απαντήσεις. Όντω έχουμε παρόμοιες απόψει. δηλαδή Κομισιόν, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Στην κυρία Χολμάγερ να πω ότι βεβαίω ο Επίτροπο, είναι πάντα έτοιμο να σας ενημερώσει. Αν δεν μπορεί να έρθει ο ίδιος, ε, έρχομαι εγώ, είμαι διαθέσιμος. Συμμερίζομαι το αίτημά σας σε σχέση με το, το, προσωπικό το έχω ήδη πει για τη Europol και τα, όσα είπατε για τα συστήματα κρυπτογράφησης. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, γιατί το έχουμε συζητήσει και στο φόρουμ ε, για το ίντερνετ, με τις εταιρείε ίντερνετ. Πρέπει να βρεθεί σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία έκφρασης και την πρόσβαση σε πληροφορίες. κόπτη ο μιλητής. Παρακαλώ. Όσον αφορά τα όσα είπε η κυρία Βερζιά, συμφωνώ μαζί σας. Θα είδατε τους τελευταίους μήνες και επίσης από την Κομισιόν ότι δεν έχουμε αντιδράσει ε, πανικόβλητη, αλλά Έχουμε μετριοπαθείς αντιδράσεις και επίσης έχουμε ε, υπογραμμίσει πολύ προσεκτικά ότι πολλές προτάσεις είναι ήδη επιτάπητος εδώ και καιρό και ότι ήδη συζητάμε. Δεν αντιδρούμε πανικόβλητη, λοιπόν. Στην κατάσταση. Αν και, και συμφωνώ με την κυρία Μόρσεν ότι μάλλον είμαστε σε διαφορετικό πλαίσιο. Το πλαίσιο έχει αλλάξει και πρέπει να το δούμε τις επόμενες εβδομάδες γιατί η γαλλική κυβέρνηση ε, έχει ενεργοποιήσει το 42.7, το άρθρο 42.7, αλλά εντός της Ένωσης αυτό δεν μας βάζει σε πολύ διαφορετική κατάσταση. Όσον αφορά το δίκτυο ΡΑΝ, κυρία Σαργεντίνη, δεν έμεινε ότι μισή μέρα στο γραφείο μου. Πρέπει να δω τι έγινε. Αλλά είμαι ευτυχής που αυτό το κέντρο αριστείας έχει δημιουργηθεί. Είναι λειτουργικό. Και όσον αφορά τους άλλους συναδέλφους, Νομίζω ότι ο κύριος Μπράουν έχει ήδη δώσει την απάντηση. Κάτι που θέλω να υπογραμμίσω δε είναι ότι για την ώρα λειτουργούμε στο πλαίσιο όσο γίνεται της ε, μεταναστευτικής κρίσης και στο λειτουργικό σύστημα Σέγγεν, αλλά πρέπει να προσέξουμε πάρα πάρα πολύ. Να μην αμφισβητηθεί το Σέγγεν. Και μια από τις βασικές συζητήσεις που θα γίνουν τις επόμενες μέρες και εβδομάδες και μάλιστα και αύριο ανάμεσα στους υπουργού Εσωτερικών θα είναι να εξετάσουμε πώς θα εξασφαλίσουμε ότι το Σέγγεν θα μπορέσει να διατηρηθεί και να εξακολουθήσει να θεωρείται ως ένα λειτουργικό σύστημα από τους Ευρωπαίους πολίτες και ίσως θα πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Μια θα είναι η πρόταση που κάνουμε ε, όσον αφορά τους ε, Ευρωπαίους συνοριοφρουρούς που θα συζητηθεί θέμα που θα συζητηθεί από το Δεκέμβριο. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Είμαστε ευγνώμονες που ήρθατε και καταλαβαίνω ότι πρέπει να φύγετε και ε, που μείνατε στη συζήτησή μας και προσπαθήσατε να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ. So, colleagues, as I enlisted the names, we have a long list. That means... Λοιπόν, έχουμε ένα μακροσκελή κατάλογο και ίσως χρειαστεί να ε, αλλάξουμε το σχεδιασμό Τη συνεδρίασής μας, θα έπρεπε να έχει ήδη τελειώσει τώρα στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν, δίνω το λόγο. Στου συντονιστέ και μετά θα χρειαστήσω και να πέμβω αν τυχόν κάποιος ξεπεράσει το χρόνο, Κύριο Κουέλιου. Ευχαριστώ. Άκουσα ότι έχουν κορεπέρ, αλλά θέλουμε να μιλήσουμε και στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Του ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Διευθυντή τη Γεροπόλη για τη δήλωση. Ήταν τραγωδία, επίθεση. Δέχτηκαν οι ίδιε οι αξίε και αρχέ μα και με, με ανησυχεί ότι άλλοι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν αυτό. Δύο πράγματα μου ανησυχούν ιδιαίτερω. Η σύνδεση που γίνεται ανάμεσα στους τρομοκράτες ε, ε, και τους πρόσφυγες, κάποιοι για δημοτικούς λόγους κάνουν αυτή την ασφαλμένη σύνδεση και το Σέγγεν επίσης ε, τίθεται εν κινδύνο που είναι σύμβολο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος για τα εσωτερικά σύνορα καταλαβαίνω ότι τα κράτη-μέλη Εάν ε, χρειαστεί, αν παραστεί ανάγκη, έχουν το δικαίωμα να επανεισάγουν ελέγχου στα σύνορα. Όμω λύση δεν είναι. Είναι προσωρινό μέτρο. Και χρειαζόμαστε περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις εθνικές αρχές και του Europol και τι υπηρεσίες πληροφοριών. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Ε, κάθε χώρα μόνη της είναι πιο αδύναμη. Πρέπει να ενωθούμε. Εάν έχουμε καλούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Κάποια κράτη-μέλη όμως έχουν ξεχάσει ότι τους αλλοδαπούς μαχητές μπορούμε να τους καταγράψουμε και να τους έχουμε υποπαρακολούθηση. Χρειαζόμαστε ανθρωπίνους πόρους περισσότερους από όλα τα κράτη-μέλη στα εξωτερικά σύνορα και καλύτερη επιμελητή. Επίσης θα πρέπει να εφαρμοστεί το νέο σύστημα πληροφοριών του Σόγγι διότι είναι ξεκάθαρα τα προβλήματα που έχουμε. Ε, σε επίπεδο ελέγχου των εξωτερικών συνόρων και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση ότι χρειαζόμαστε ελευθερία μετακίνησης, αλλά χρειαζόμαστε και ασφάλεια. Σας ευχαριστούμε, Λόπες Αγγιλά. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστώ και τον κύριο Ράιτ ε, που μένει αντίθετα από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπή. Και στην πραγματικότητα αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το δυναμικό που έχει η Europol για πρόοδο προς ε, αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών που δεν υπάρχει. Υπάρχει σε εμβριακή μορφή με μια σειρά κεφαλαίων που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας για την πολιτική ασφάλειας, άμυνας, ολοκληρωμένη διαχείριση εξωτερικών συνόρων. Όλα αυτά είναι σχετικά. Αλλά το δυναμικό της ανάπτυξης μιας πραγματικής μονάδας, ευρωπαϊκής μονάδας πληροφοριών, τι θα ήταν, τι όραμα έχετε εσείς κύριε Wainwright για την εξασφάλιση της λειτουργίας ενός ΣΙΤΣΕΝ, ενός κέντρου αναλύσεως καταστάσεων, Situation Center, με αναλυτές. Ε, και προσωπικό από τα διάφορα κράτη-μέλη, γιατί το δεδομένο ότι μπόρεσαν οι τρομοκράτες που διέφυγαν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι να ξεφύγουν παρότι τους είχαν ελέγξει οι γαλλικές αρχές από τον έλεγχο των βελγικών αρχών και να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο στην πόλη που γεννήθηκαν, δηλαδή τις Βρυξέλλες, είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Θα ήθελα λοιπόν πιο, πολύ, πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Έχουμε εστιαστεί στην επίδειξη αλληλεγγύης, συμπόνιας, ενσυναίσθησης σε σχέση με τα θύματα και τους εκείνους τους, αλλά ίσως πρέπει να κοιτάξουμε και περαιτέρω τους κινδύνους που απειλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις και σε αυτούς που θέλουν μια πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση και σε εκείνους που θέλουν μια πιο εθνική προσέγγιση και σε αυτούς που θέλουν να κάνουν αμάλγαματα μεταξύ, να αναμίξουν την πολιτική αντιμετώπιση τρομοκρατίας με τη μεταναστευτική πολιτική και το άσυλο. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να μας δώσει απαντήσεις η Europol. Ευχαριστώ. 11 μήνε μετά το ροσαλή Επτό πρέπει να περάσουμε στις πράξεις και να δώσουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση ε, στον πόλεμο που έχει ξεκινήσει η Αλταές ε, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στην Ευρώπη. Ας ξεκινήσουμε με τις ρίζες του κακού και όπως είπε ο εκπρόσωπος της Λουξεβουριανής Προεδρίας, ένα βασικό θέμα είναι η χρηματοδότηση. Το Ισλαμικό κράτος ε, με τις πετρελοπηγές της Συρίας και του Ιράκ και με αυτούς που δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι, δεν θα τους κατονομάσω, αλλά ξέρουμε όλοι περί τίνος πρόκειται, που τους εξασφαλίζουν χρήματα, ε, εξασφάλισαν χρηματοδότηση. Πρέπει να στεγνώσουμε το Ισλαμικό κράτος από κονδύλια. Ε, τώρα υπάρχει το θέμα της στρατιωτικής παρέμβασης, δεν είναι θέμα της ε, ΛΥΜΠΕ, αλλά η Γαλλία συμμετέχει στις ε, επιθέσεις κατά των πετρελαιοπηγών. Τώρα, όταν μιλάμε για λοδαπούς μαχητές, μα τι οι Ευρωπαίοι μαχητές, πρέπει να τους ονομάζουμε Ευρωπαίους μαχητές, περνούν από διάφορα αεροδρόμια από τη Συρία και έρχονται στην Ευρώπη. Στη Λιμπερασιόν σήμερα το πρωί αναφερόταν ότι υπάρχουν Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ε, αεροδρομίων στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα, στην ε, Τσεχία, στην Εστονία και στην Ουγγαρία που είναι αρκετά ανοιχτά ώστε να μπορούν να περνούν άνετα οι, αυτοί οι Ευρωπαίοι μαχητές. Ε, για τον τριμερή διάλογο θα πρέπει να ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος του 2015 όλα και τα τρία θεσμικά όργανα έχουν αναλάβει δέσμευση για αυτό, για την ανταλλαγή τώρα πληροφοριών χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα ότι θα έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας ε, κύριε Wainwright και πάλι εδώ να περάσουμε στις πράξεις ε, γιατί πολλά ακούμε, πολλά λέμε και από τον κύριο Μπριζάρ που είναι ο, ο διευθυντής του Γαλλικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας ε, όμως το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ε, συνεργασία χωλένουμε στην ανταλλαγή πληροφοριών να δράσουμε Ευχαριστούμε. Γιγιόμ. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά που ακούσαμε ήδη. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για την, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και την συμπόνια μου προς τα, τις οικογένειες των θυμάτων. Για να προχωρήσουμε όμως να πω ότι ε, δέχθηκε το πλήγμα η Γαλλία, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα οποιοδήποτε όλοι απειλούνται. Άρα τίθεται το ζήτημα της αλληλεγγύης. Τι κάνουμε, ε, πώς μπορούμε να ανασχηματίσουμε τις ε, διπλωματικές σχέσεις μας με τις χώρες της περιοχής, σε τι εικόνα προβάλλουμε σε διεθνές επίπεδο, ε, ένοπλη παρέμβαση μας επικαλέστηκε το άρθρο 42.7 ο πρόεδρος για την στρατιωτική αλληλεγγύη, πέραν αυτού έχουμε και την οικονομική αλληλεγγύη όχι μόνο για αυτούς που θα χρειαστούμε για την επέμβαση την ίδια, αλλά ε, και για την παρακολούθηση, για την εποπτεία της κατάστασης, για την πρόληψη. Η αλληλεγγύη σε όλες τις εκφάσεις της είναι σημαντική. Είπατε ότι το Συμβούλιο την Παρασκευή θα ασχοληθεί με διάφορες πτυχές του ζητήματος ε, και ακριβώς αυτό ήθελα και εγώ, διότι φοβάμαι ε, ότι δεν θα μιλήσουμε για το ζήτημα της ανταλλαγής πληροφοριών, γιατί είπαμε πολύ πολλοί δεν είναι ικανοποιητικός ο και θα πρέπει να βαθμιστεί έλεγχος ε, των όπλων, ρίζοσπαστικοποίηση, φοβούμουν ότι θα αποσιωπούνταν αυτά τα ζητήματα, αλλά και το θέμα PNR δεν είναι πανάκια, δηλαδή χρειαζόμαστε το πακέτο, χρειαζόμαστε ολόκληρη εργαλειοθήκη. Κάθε θέμα ξεχωριστά δεν ε, επαρκεί. Ε, ε, εξάλλου αυτή την εντολή έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συνολικό πακέτο για την εργαλειοθήκη. Θα ήθελα να μιλήσω για την ε, συνολική δέσμευση ως προς ε, την πρόληψη, ένα βασικό ζήτημα Όντως χρειαζόμαστε πιο εξισορροπημένες σχέσεις με τις χώρες στην περιοχή για την αναπτυξιακή βοήθεια μέσω μακροπρόθεσμα αν θέλουμε να αλλάξουμε τις σχέσεις που έχουμε με τις χώρες αυτές γιατί από αυτούς προέρχονται οι άνθρωποι που τελικά οργανώνουν θερμοκρατικές επιθέσεις. Και μην ξεχνάμε ότι οι νέοι Ευρωπαίοι ε, σκότωσαν, δολοφόνησαν άλλους νέους Ευρωπαίους σε θέματα πρόληψη λοιπόν και θέματα ευθύνης. Ε, μίλησα εδώ με κάποιους που ασχολούνται με την υποδοχή των των μεταναστών και τελικά ε, ε, ε, ανακάλυψαν τη δεσμευσή τους μας. Πώς, πώς μπορούν να εξομοιώνουν τους εγκληματίες με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που προσπαθούν να ξεφύγουν από το Ισλαμικό κράτος. Θα τους ρίξουμε στην αγκαλιά τους μέσα αν τους γυρίσουμε την πλάτη. Ευχαριστώ, Αναγκόμες. Θέλω να πω ότι η επίθεση στρέφεται εναντίον όλων μας και το ξέραμε ότι θα λάβει χώρα. Το είπε και ο κύριος Βουέινραιτ ότι ήταν αναμενόμενοι και αναμένονται και επόμενες. Είναι λοιπόν εξωφρενικό το ότι δεν έκαναν τα κράτη-μέλη αυτό που όφυλαν να κάνουν. Και το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να απαλλαγούμε από τις ηλίθιες οικονομικές πολιτικές οι οποίες ε, τροφοδοτούν τον κοινωνικό αποκλεισμό και κυρίως τους μετανάστες δεύτερης γενεάς αυτούς, δηλαδή από την ε, ομάδα των οποίων προέρχονται οι τρομοκράτες και δεν είναι ξένοι. Οι τρομοκράτες είναι Ευρωπαίοι. Ερωτώ λοιπόν κύριε Wainwright πόσα αξιολογείται τα προγράμματα πρόληψης της ε, ριζοσπαστικοποίηση, ιδίω σε επίπεδο φυλακών που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουν υλοποιήσει τα κράτη-μέλη, αλλά δεν ε, υλοποίησαν γιατί μεταξύ άλλων δεν είχαν τα χρήματα που απαιτούνταν. Άλλο ζήτημα βεβαίως είναι αυτό των ε, εφιών συνόρων, smart borders είναι ευφυές το να μην ανοίγουν ασφαλείς και νόμοι δρόμοι για τον μετανάστη ώστε να περνάει μέσα από έναν έλεγχο τακτικό και ε, κανονικό είναι ευφυές το να αμφισβητείτε το ίδιο το Σέγγεν, γιατί γνωρίζουμε ότι όταν δεν υπήρχε το Σέγγεν από την πατρίδα μου, την Πορτογαλία, πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες έφυγαν για να φτάσουν στη Γαλλία και τη Γερμανία, περνώντας φυσικά παράνομα τα σύνορα. όταν είχαμε το Σέγγεν, λέει ο Μιλήτρια. Το PNR, το σύστημα ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Βεβαίω, είναι ένα εργαλείο, το έχουμε και σαν ε, πρόταση για εγκρίση την προηγούμενη εβδομάδα για την αποφυγή και την αποτροπή τη ριζοσπαστικοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο, όπω είπε ο κύριο Μπράουν, θα το ε, προβάλλουμε σαν ε, απάντηση στους πολίτες. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικά εργαλεία, αποτελεσματικά εργαλεία που σημαίνουν πλήρως προσαρμοσμένα στην προστασία των δεδομένων. Και εκεί πρέπει να κάνουν κάποιες κινήσεις τόσο η Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο και όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε και θα είμαστε παρόντες στη συζήτηση. Όπλα, τα κράτη-μέλη δεν υλοποιούν προφανέστατα, την κοινή θέση για τις εξαγωγές των όπλων και δεν εξάγουν το εμπόριο των όπλων μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων. Για να μην μιλήσω για κάποιες χώρες οι οποίες έφτασαν να κάνουν και πληστηριασμούς όπλων μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι. Σέγγεν λοιπόν. Και είπε ο κύριος Ρούτε να κάνουμε αυτό που λέμε και να δώσουμε τα χρήματα που απαιτούνται για να ελοπίσουμε τις προσχέσεις μας. Προσωπικό, δυναμικό, δυνατότητες, ε, ανταλλαγή πληροφοριών, UIFs, ε, αστυνομία. Για να πάμε να δούμε πού είναι αυτοί οι υπάλληλοι ε, στα κράτη-μέλη έχουν τον εξοπλισμό. Υπάρχουν αυτές οι μονάδες οι ειδικέ έχουν εξοπλισμό, έχουν επικοινωνία με τα κέντρα της Europol. Βεβαίως το ίντερνετ είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε υποστηρίξει την πρόταση αυτή, την έχουμε γράψει στην, έκθεσή μας. Δεν, δεν εμποδίζει την υλοποίηση αυτής της λύσης στο Κοινοβούλιο, αλλά κάποια άλλη. Κυρία Σουινμπέρν. Ευχαριστώ. Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη στην, ε, στο Παρίσι. Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψουμε ότι υπάρχουν κάποιοι εδώ στις ευρωπαϊκές χώρες ε, ε, που πίστεψαν αυτούς τους ανθρώπους ε, και τελικά έχει βγάλει ρίζες το ριζοσπαστικό Ισλάμ εδώ στις δικές μας κοινωνίες και βλέπουμε τι συνέβη με την ελεύθερη μετακίνηση και της ανύπαρκτης ουσιαστικά προστασίας. Βλέπετε ποια κατάσταση έχει δημιουργηθεί γιατί ο Προφρόντεξ είχε ασχοληθεί με την προστασία των συνόρων. Όμως το 98% των κονδυλίων τα διοχετεύουν σε έρευνα και διάσωση, σε τέτοιες επιχειρήσεις. Ποιο προστατεύει τα δικά μας τα σύνορα, κανεί μπαίνουν όπλα, ναρκωτικά, ε, τρομοκράτες, ε, είναι διάτρητα τα σύνορα, δεν υπάρχει πουθενά έλεγχος. Ε, ποιος την έχει φτιάξει αυτή την κατάσταση, πώς καταλήξαμε σε αυτή την κατάσταση που είναι απειλή για την ασφάλεια των ίδιων των πολίτων. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να τους απειλήσουμε με, τα ίδια όπλα να τους πολεμήσουμε, να πολεμήσουμε αυτούς τους δολοφόνους και τους τρομοκράτες και βιαστές. Αντί να κάνουμε αυτό, τους λέμε, σκεφτόμαστε πώς να τους ενσωματώσουμε στις κοινωνίες μας. Ε, δηλαδή, τι θέλουμε να τους δώσουμε και θέση στην αγορά εργασίας. Ε, είναι δολοφόνοι, δεν μπορώ, δηλαδή, τι να πω πια. Είναι αποβράσματα αυτοί οι άνθρωποι και μπαίνουν στις, ε, στις χώρες μας δίπλα στους φιλήσυχους πολίτες. Ε, ε, όταν πηγαίνουν στη Συρία δεν πρέπει ποτέ να τους επιτρέψουμε να ξανάρθουν, να μην ξαναπατήσουν το πόδι τους εδώ πέρα. Δεν μπορώ να νιώσω ασφάλεια όταν ξέρω ότι επιστρέφουν αυτοί οι άνθρωποι. Ο θαλμός αντί οφθαλμού Με τα ίδια όπλα θα πρέπει να τους πολεμήσουμε και να αποτρέψουμε έτσι την περαιτέρω προσαστικοποίηση. Ευχαριστούμε. Ε, Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι ε, είναι φοβερές αυτές οι επιθέσεις και θα πρέπει να προβληματιστούμε και να αντιδράσουμε σωστά ε, επιδιώκοντας περισσότερη ασφάλεια αλλά διαφυλάττοντας και τον τρόπο ζωής που δέχεται επίθεση. Δεν νομίζω ότι ήρθε η ώρα τώρα να ζητήσουμε υιοθέτηση μέτρων που δεν καθίστανται αναγκαία μετά από τις ε, επιθέσεις, υπερβολικά μέτρα. Θα πρέπει να προβληματιστούμε για τη συνέχεια. Ε, ξέρετε, βρήκα λίγο ανάρμοστα τα σχόλια του κυρίου Ρούτε για την κρυπτογράφηση. Δεν υπάρχει ε, με ενδιάμεση κατάσταση, είτε είστε υπέρ είτε κατά της κρυπτογράφησης και ε, για την μυστικότητα των επικοινωνιών, για την ηλεκτρονική επικοινωνία Είμαι κατά. Ε, δεν, ε, η, η μυστικότητα των επικοινωνιών ε, συνιστά επίσης δικαίωμα δίπλα στην ελευθερία έκφρασης στη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πώς μπορούμε να έχουμε αυξημένη ασφάλεια. Τίθεται αυτό το ζήτημα και οι τρομοκράτες προσπαθούν να παρακάμψουν τις ε, υποκλοπές, ε, χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας. Εξ αρχής ήταν ξεκάθαρο, ακόμη και με κρυπτογράφηση, πάντοτε υπάρχουν πληροφορίες ε, για το συντονισμό των τρομοκρατικών ενεργειών και εμείς μπορούμε ε, να ε, έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Γιατί δεν μίλησε για, τα κοινά για τις κοινέ ερευνητικές ομάδες ο κύριος Ρούτε με τη Europol και Eurojust μετά το 2011 αυτή ήταν η αντίδραση που είχαμε και με αναλογικό τρόπο τα κονδύλια και οι ανθρώπινοι πόροι ε, που επενδύσαμε οδήγησαν σε ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές των κρατών μελών. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε και όχι να προσπαθούμε να βρούμε κάτι καινούργιο που δεν έχει αποδεδειγμένα λειτουργήσει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, λέει ο κύριος σεμέλο τον κύριο Βένερ Ράιτ διότι ε, παρέμεινε και δείχνω ότι σέβεται την Επιτροπή μας ε, και αυτό που θέλουμε να μάθουμε και είναι θεμητό. Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τη Γαλλία, τους Γάλλους αλλά και προς ολόκληρη την Ευρώπη γιατί ε, είχαμε και θύματα από διάφορες χώρες και Πορτογάλους. Με βάρβαρο τρόπο τους δολοφόνησαν όλοι από κοινού καταπολεμούμε την τρομοκρατία. Δεν γίνεται όμως με, ρομαντισμό να το καταπολεμήσουμε. Ε, μπροστά στον τρόμο ε, δεν μπορούμε εμείς να προτάσουμε τις αρχές μας. Πρέπει να κάτι να κάνουμε. Ε, να τους εξουδετερώσουμε. Διότι μόνο έτσι θα διαφυλάξουμε τον τρόπο ζωή μας. Θα ήθελα ένα συγκεκριμένο ερώτημα να θέσω, διότι... Ε, εγώ ξέρω ότι οι τρομοκράτες ε, δεν είναι πρόσφυγες. Ε, κάνω τη διάκριση. Γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ευρώπη. Είναι τρομοκράτες όμως. Αυτό αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις μαζικές δροές προσφύγων οι τρομοκράτες για να μπουν και εκείνοι στην Ευρώπη. Οπότε, γι' αυτό το λόγο θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Στο κέντρο στα κέντρα υποδοχής προσφύγων θα ε, πρέπει να προσέξουμε να μην ε, έχουμε ε, δούριους ύπους που θα επιτρέψουν να, στους πρόσφυγες να μπουν έκνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε γύρω στους 4.000 αλλοδαποί μαχητές, λέει ο Ίσης, μπαίνουν, έχουν μπει στην Ευρώπη μέσα από αυτά τα κέντρα υποδοχής. Αυτό προκύπτει από στατιστικές του Ερευνητικού Ινστιτούτου της Ρωσίας γιατί και εκείνοι επλήγησαν έτσι ολόκληρο αεροσκάφος κατερρευθεί και ήταν πάρα πολλά τα θύματα της ε, τρομοκρατικής επίθεσης. Ο διευθυντής αυτού του Ινστιτούτου λέει λοιπόν ότι είναι μια υπαρκτή απειλή 4.000 ε, μαχητές ε, που μπορεί ήδη να έχουν μπει ήδη στην Ευρώπη. Πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά αυτό τον ισχυρισμό πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά ότι χρησιμοποιούν τα κέντρα υποδοχής οι τρομοκράτες για να μπουν στην Ευρώπη. Ευχαριστώ.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 Πρόκειται για τραγικά γεγονότα και δεν μπορούμε να τα αντιπαρέλθουμε, θα πρέπει να αντιδράσουμε με κάποιο τρόπο. Δυστυχώς ε, φοβάμαι ότι μπορεί συχνά από εδώ και πέρα να ζούμε τέτοια περιστατικά, οπότε με σύνεση θα πρέπει να αντιλήσουμε τα συμπεράσματα με συστηματικό τρόπο, ε, να αντιδράσουμε με συνέπεια και να είμαστε και αποτελεσματικοί τον τρόπο που αντιδρούμε. Είναι σημαντικό ε, σε αυτή τη συζήτηση να κάνουμε ε, εντατικά τις ανταλλαγές απόψεων με τους εκπροσώπους των αρμοδίων ε, οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά τώρα το να αντιδράσουμε με σπουδή προκύπτει από την ανάγκη ε, γρήγορη αντίδραση ε, σε, αυτά τα περιστατικά. Όντω πρέπει να δράσουμε με σπουδή, αλλά ταυτόχρονα με λογή. Ε, προέκυψε στη συζήτηση το θέμα των ευφυών συνόρων και Ποιο είναι το ζήτημα να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις εισόδους, ε, να ελέγξουμε και τις εισόδους των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και μέσα σε αυτή την ε, σπουδή και τη δυναμική μετά τα περιστατικά προτείνονται ίσως υπερβολικά εσπεσμένα μέτρα. Θα πρέπει όμως να τα συζητήσουμε Ε, γιατί θεωρώ ότι ο περιορισμός της ελεύθερης μετακίνησης ε, μπορεί να οδηγεί σε περιορισμό της ε, ασφάλειας. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα συστηματικό τρόπο προσέγγισης του ζητήματος. Ευχαριστούμε κύριος Γιούρακ. Ε, είχα την εντύπωση ότι ε, δέχτηκε η δική μου η χώρα επίθεση όταν έβλεπα τις τρομοκρατικές ε, επιθέσεις και θα πρέπει να διαπιστώσουμε ποια είναι η ευρύτερη σημασία αυτών των περιστατικών. Με ακούτε? Ναι. Δεν υπάρχει η μετάφραση. Όχι. Θα τα ξαναπώ. Μετά τις επιθέσεις της Παρασκευής ε, είχα την εντύπωση ότι όλα είχαν συμβεί στη χώρα μου. Ε, πρόκειται όμως δυστυχώς για την αρχή μια σειρά επιθέσεων. Ε, δεν ε, είναι μια άπαξ τραγωδία, διότι πέρα από τη Μέση Ανατολή επιτίθεται και εδώ το Ισλαμικό κράτος και θα πρέπει να αναμένουμε και άλλες τέτοιες επιθέσεις. Αυτή η σειρά δημοκρατικών επιθέσεων δείχνει πως έχουμε να κάνουμε με, μια οργάνωση που είναι αποφασισμένη να συνταράξει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσοι μαχητές ε, του Ισλαμικού κράτους έχουν μπει στην Ευρώπη, αναρωτιόμαστε. Εγώ θα αναρωτηθώ κάτι άλλο. Ποια είναι η κοινωνική βάση αυτών των δραστηριοτήτων, αυτών σε ποιο βαθμό δέχεται υποστήριξη του Ισλαμικού κράτους επί τόπου. Δηλαδή, σε πόσα τζαμιά, σε πόσους τόπους λατρείας υποστηρίζονται ή αντίστοιχα, αντίθετα μάλλον απορρίπτονται οι δραστηριότητες ε, αυτές. Ε, ποιος συμμετέχει στην προπαγάνδα του Ισλαμικού κράτους, ε, ποιος Ποιος μπορεί να λειτουργεί ως κοινωνικό έρισμα ε, αυτών των ε, τρομοκρατών. Ποιοι είναι οι υποστηρικτές τους. Ποιοι εγκρίνουν ε, τη δράση τους. Τον Απρίλιο αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πως πρέπει να καταπολεμήσουμε τους διακινητές και την παράνομη μετανάστευση. Αυτή η επιχείρηση Σοφία. Σοφία. Η... Έχει ξεκινήσει και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όμως με τόσο περιορισμένου εύρους ε, επιχειρήσεις ε, το μεγάλο ε, αριθμό σκαφών που φτάνουν στις ακτές μας. Ευχαριστώ η Κορνέλια Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ε, προσθέσω, δεν θέλω να προσθέσω κάτι, τα είπε ο συνάδελφος, θα ήθελα μόνο να θέσω κάποια ε, ερωτήματα. Ε, ε, αναρωτιέμαι σήμερα μήπως οι Υπουργοί Οικονομικών θα έπρεπε να ασχοληθούν και με τις οικονομικές τροές για να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις μεταφορές χρημάτων προς τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτό θα με ενδιέφερε. Θα έπρεπε λοιπόν να συζητήσουν ε, μήπως ε, δεν έπρεπε να επιτρέψουν καμία εξαγωγή όπλων προς τη Μέση Ανατολή. Όμως ε, αυτά συμβαίνουν, εξακολουθούν να συμβαίνουν και μην ξεχνάμε ότι το, στο Ιράκ μεγάλος ο στρατός με αμερικανικά όπλα γιατί τα άφησαν οι Αμερικανοί φεύγοντας στο Ιράκ τα όπλα και σήμερα αυτή είναι η βάση της κατάστασης. Γι' αυτό στη Συρία έχει ανθίσει τόσο πολύ η τρομοκρατία και ε, ε, έχουμε αυτά, αυτές τις θλιβερές ε, τρομοκρατικές επιθέσεις. Κύριε Ρόιτε, έχουμε στη Γαλλία σύστημα PNR. Ένα εκατομμύριο επιβάτες πέρσι καταχωρίστηκαν βάσει αυτού του συστήματος PNR. Μα τι λέμε τώρα, χρειαζόμαστε κι άλλα πρέπει να ε, αναπτυχθεί περαιτέρω το σύστημα PNR. Και κάτι άλλο για το Frontex. <laughs> Είπατε εσείς πως, ε, μάλλον ο πρέσβης Μπράουν το είπε, ο Frontex μαζί με τη Europol πρέπει να καταπολεμήσουν από κοινού το εμπόριο όπλων. Mm πώς το έχουμε φανταστεί, θα θα ε, κάνετε κάτι καινούριο, ε, δηλαδή δεν το κάνει ήδη ο Frontex αυτό, αυτό θέλετε να μας πείτε. Ε, και νομίζω ότι θα έπρεπε να αναρωτηθούμε για κάποια λεπτά με ποιο τρόπο στη Γαλλία και στην Ευρώπη γενικότερα μπορούμε να προλαμβάνουμε την ριζοσπαστικοποίηση αντί να διορθώνουμε τα κακό σκήμενα όταν προκύπτουν. Now I give back the floor to uh, Mr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 Προεδρείου μονάχος. Θα προσπαθήσω όμως να απαντήσω. Ο κύριος Λόπες Αγιράρ ε, μίλησε για μια μελλοντική ενδεχόμενη υπηρεσία πληροφοριών για την Ευρώπη. Εσείς είμαστε ρεαλιστές όμως για το ποιο θα μπορούσε να είναι το επίπεδο πολιτικής αποδοχής για ένα τέτοιο εγχείρημα. Ξέρετε ότι η συνθήκη ορίζει ως αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ως εκ τούτου της ε, υπηρεσίας πληροφοριών. Δεν υπάρχουν τους ή άλλως λειτουργικές εξουσίες, μόνο πολύ καλή δουλειά που μπορεί να γίνεται ασφαλώς, αλλά ε, εστιάζεται κυρίως στην ανταλλαγή στρατηγικών πληροφοριών, εκθέσεων ε, αξιολόγησης, που δεν μπορούν όμως να θεωρηθούν ως μια υπηρεσία πληροφοριών, αυτό που κάνει η Europol. Υποστηρίζουμε το λειτουργικό έργο και με αυτή την ε, δράση της υποστήριξης πρέπει να πω ότι δεν μπορούμε να θεωρηθούμε ως FBI ότι έχουμε κάποια εκτελεστική εξουσία η επιβολή της τάξης. Μια κοινή πλατφόρμα μπορούμε να προσφέρουμε, μια κοινή ευρωπαϊκή πλατφόρμα για ανταλλαγή των πληροφοριών. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο όλο και περισσότερο, καθώ είναι διεθνεί διαστάσει τη τρομοκρατία αλλά και του οργανωμένου εγκλήματο. Χωρί λοιπόν αρμοδιότητε, ακόμη και χωρί αρμοδιότητε επιβολή του νόμου, η Europol μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο. Και αυτό μέχρι ότου εκδηλωθεί και η πολιτική βούληση, η ανοίξη, η πολιτική όρεξη για κάτι περισσότερο. Ε, τώρα γιατί η ανταλλαγή των πληροφοριών δεν είναι ήδη καλύτερη μεταξύ των υπηρεσιών. Αυτό το ρωτήσατε πολύ. Το ζήτημα είναι ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών μελών και νομίζω ότι η ανταλλαγή των πληροφοριών έχει σημαντικά βελτιωθεί και είναι αρκετά αποτελεσματική ε, μεταξύ υπηρεσιών πληροφοριών. Από την άλλη, η ανταλλαγή συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών αρχών έχει βελτιωθεί και εκείνη από πλευράς της. Εγώ όμως θέλω ιδιαίτερα να εστιαστώ στην ανάγκη για διασύνδεση της δουλειάς συλλογή πληροφοριών και της αστυνομικής δουλειάς που πρέπει να εξασφαλίσει η Europol. Αυτή είναι η δουλειά μας για να, έχουμε πιο να εξασφαλίσουμε μια πιο αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και όπως είπα και νωρίτερα αυτό κυρίως στο πλαίσιο των όσων αποτελούν μια σαφή απειλή την διασύνδεση μεταξύ εγκλήματος τρομοκρατίας, αστυνομικών ερευνών, υπηρεσιών πληροφοριών. Αυτό προσπαθούμε ακριβώς να χτίσουμε. Μια καλύτερη πλατφόρμα δηλαδή να προσφέρουμε και αυτό με την αναβάθμιση των πρωτοκόλων ασφαλείας, με πιο συχνή επικοινωνία με τις υπηρεσίες πληροφοριών. Αλλά και πάλι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και αρμοδιότητα δική τους να αποφασίσουν πόσες πληροφορίες θα διαθέσουν μέσω της Europol. Αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε αύριο για τα εξωτερικά σύνορα και Βεβαίως το ζήτημα το σχετικό με την τρομοκρατία και τη μετανάστευση. Από αστυνομικής ε, προοπτικής μπορώ να σας πω ότι χρειάζεται να γίνει βελτίωση των ε, ε, της διάγνωσης ενδεχόμενου κινδύνου ασφαλείας κατά την ε, διέλευση των συνόρων. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα και αποτελεσματική δυνατότητα διάβασης για τους μετανάστες, αλλά και ταυτόχρονα διάγνωση αποτελεσματική όποιου προσπαθεί αφικνούμενος ε, να προχωρήσει σε εγκληματικές δραστηριότητες, όποιες και είναι αυτές και πρέπει να είμαστε θέσει να κάνουμε τη διάκριση χωρίς να υπονομεύουμε βεβαίως την ε, όλη ανάγκη για διευκόλυνση κατά τρόπο αποτελεσματικό της κρίση μετανάστευση Η Europol για την ερώτηση του κυρίου και ο ρόλο της Europol στα σύνορα. Είναι κατά κύριο λόγο να εντοπίσουμε τους λάθροδιακινητές, τα σχετικά δίκτυα, την, τα δίκτυα εκμετάλλευσης των μεταναστών με την παροχή παράνομων ε, υπηρεσιών και έτσι έχουμε την επικοινωνία με τους ε, συναδέλφους που εργάζονται στον χώρο των συνοριακής φύλαξης. Τώρα πρέπει να ξανακοιτάξουμε αν είναι σε θέση η Europol να υποστηρίξει μια ευρύτερη ε, δράση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται τώρα. Πρέπει λοιπόν να έχει μια αποτελεσματική διάγνωση τρομοκρατικού, ε, ε, συγγνώμη, κινδύνου για την ασφάλεια γενικά συνεργασία με χώρες της περιοχής της ευρύτερης περιφέρειας. Πολύ σωστά υπόθηκε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μας ε, με χώρες της περιοχής. Αυτό είναι η κίνηση βεβαίως που θα πρέπει να κάνει και η Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η Europol Υπηρεσίες προσφέρει μόνο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε, μια, σε έναν πιο αποτελεσματικό διάλογο και συνεργασία με τις ανλόγω λόγω χώρες στο εγγύς μέλλον. Έχουμε σοβαρές ανησυχίες σε σχέση με την ε, με τις δυσφαλιστικές δικλείδες ασφάλειας ε, δεδομένων που θα χρειαστεί να διαθέσουμε στις χώρες της περιοχής, αλλά υπάρχει σαφώς ενδιαφέρον για ανταλλαγή και πάνω απ' όλα αποδοχή από πλευράς της Europol προσωπικών δεδομένων για άτομα επικίνδυνα που μπορούν να αποτελούν ε, κίνδυνο ασφαλείας, αλλά και εμείς θέλουμε αυτό να το πράξουμε πάντα με σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των δικών μας πολιτών σε σχέση με τις χώρες αυτές και είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει και να βρούμε λύσεις. Η κυρία Γκόμες που με ρώτησε για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης. Μάλλον δεν είμαι ο καταλληλότερος να σας δώσω την τέλεια απάντηση. Μπορώ όμω να μιλήσω για την εμπλοκή των αστυνομικών αρχών και ιδιαίτερω τη Europol στην προσπάθεια αυτή που προσπαθεί στοχευμένα να καταπολεμήσει τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται το ίντερνετ ως μείζον παράγων της από τους εγκληματίε αυτούς. Σημαντικός, τεράστιο θα έλεγα όγκο, υλικού, προπαγανδιστικού εργαλείου δηλαδή, περνάει μέσα από το ίντερνετ και έχουμε μια μονάδα, την Internet Referral Unit, η οποία καθημερινά διαχειρίζεται τεράστιο όγκο περιπτώσεων, προσπαθώντας να αποτρέψει την ISIS από το να χειραγωγήσει αυτό το κομμάτι των ελευθεριών που έχουμε εξασφαλίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να... και να, το... να τις αξιοποιήσει για το βρώμικο αυτό εμπόριο ψυχών. Επίσης, Θα ήθελα να αναφέρω επίσης ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για πιο αποτελεσματική συνεργασία σε επίπεδο και κρατών μελών και με συμμετοχή της Eurojust. Αυτό θα σήμαινε προ ε, εμφάνιση ενώπιον του δικαστή, συνεργασία, δηλαδή εντοπισμό, διασύνδεση σε λειτουργικό επίπεδο, σε επιχειρησιακό επίπεδο καλύτερα και μεικτές ομάδες με τη Eurojust. Για την κυρία Ernst, πληροφορίε για τι οικονομικέ κινήσει. Συμφωνώ απολύτω. Θα πρέπει οι προσπάθειέ μα να ενισχυθούν στο με αυτόν. Εισαγωγικά και εγώ σα είπα για τι ομάδε μα ε, TFTP ε, για τον επόμενο χρόνο και στο πλαίσιο της λειτουργίας του νέου κέντρου καταπολέμησης της ε, τρομοκρατίας έχουμε μια νέα μονάδα που ονομάζεται FI Unit, δηλαδή Financial Intelligence, πληροφορίες για οικονομική δραστηριότητα και θα λειτουργήσει και αυτή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη για το οποίο και την τελεγεί των προσωπικών δεδομένων ή προσδοκίες από τα κράτη-μέλη και υποστηρίζουν βέβαια και υποστηρίζει και η Europol είναι να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα PNR συλλογή προσωπικών δεδομένων που να μπορούμε με βάση πολύ στοχευμένο ε, αντικείμενο να διαχειριζόμαστε και δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο γιατί είναι θέματα των κρατών μελών. Για τη Frontex, ε, νωρίτερα αναφέρθηκα στον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε στο, στα σύνορα. Έχουμε διακεκριμένα καθήκοντα βεβαίως και αρμοδιότητες. Έχουμε συνεργασία στο βαθμό που μπορούμε περιορισμένα γιατί δεν έχουμε ακόμα εξασφαλίσει τη συμφωνία συνεργασίας που θα μας επέτρεπε να έχουμε μια ε, τακτική ανταλλαγή και ροή προσωπικών δεδομένων από τη Frontex στη Europol. Προσπαθούμε να οδηγηθούμε στην ολοκλήρωση. Περιμένουμε από τη Frontex τελικές προτάσεις. Η Europol είναι έτοιμη από πλευρά τη. Αυτό σημαίνει τελική επαλήθευση από το EDPS, ιστορικά συστήματα σε τεχνικό επίπεδο που έχει αναπτύξει η Frontex πρέπει ακόμη να προχωρήσουν. Ίσως να μην έχουμε έχω απαντήσει σε κάθε λεπτομέρεια και σε κάθε ερώτησή σας. Ζητώ συγγνώμη, αλλά αυτά είχα να πω προς το παρόν. Και αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Μέλο που τον ξέχασα πριν, για τους πρόσφυγες και τη δυνατότητα για τους 4.000 τρομοκράτες ε, να περασ... Ναι, ευχαριστώ κύριε Μέλο και με συγχωρείτε που λησμόνησα αυτό το, αυτή την ερώτηση. Τέτοιο νούμερο εγώ δεν έχω, δεν ξέρω από πού το έχετε εσείς. Είπα εισαγωγικά ότι μας ανησυχεί ιδιαίτερος και βεβαίως ε, το λέμε, ε, μας ανησυχούν τα όσα συνέβησαν στο Παρίσι, αλλά ασφαλώς μας ανησυχούν και οι δυνατότητες για κάποιους να εκμεταλλευτούν αυτήν την κρίση, τη μεταναστευτική. Ίσως λοιπόν ε, θα ήταν καλό να μην ε, δεχθούμε αυτή την προσπάθεια να επηρεαστούμε ως προς την αποδοχή της ιδέας της μετανάστευσης. Υπάρχει μια προσπάθεια χειραγώγησης προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή να στρεβλωθεί η πολιτική για τη μετανάστευση. Αν δεν τα κάνει αυτά το ΙΚΙΛ, ακολουθούμε πληροφορίες των γαλλικών ερευνητικών αρχών και παραπάνω δεν μπορώ να σας πω στο στάδιο αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Wainwright, πληροφορίες μας δώσατε, με υπομονή μας απαντήσατε και αγαπητοί συναδελφοί ευχαριστώ για την εντατική συνεργασία στη συζήτηση αυτή. Τώρα πρέπει να δώσω πληροφορίες και είναι η εξή ότι θα αναβληθεί η συζήτηση του τελευταίου σημείου της ημερήσια διάταξης. Περνάμε στα επόμενα δύο σημεία, 7 και 8 μαζί. Μετανάστευση. Κύριε Γουένραιτ, σας ευχαριστώ και πάλι. In the context of the strategic own initiative report... Στο πλαίσιο της, ιδέας, της εκθέσεως πρωτοβουλίας για τη στρατηγική για τη μετανάστευση και τη Μεσόγειο, η κυρία Μετσόλα και η κυρία Κέγκε που δεν είναι εδώ δυστυχώς σήμερα και οι σκιωδησηγητές ε, Σπινέλη και Κοράο θα κάνουν την παρουσίαση για το έργο για το έγγραφο εργασίας για την μετανάστευση και ανάπτυξη. Σας καλώ επίσης να συστήσουμε και το σημείο 7 με την έκθεση της πρωτοβουλίας για τη μετανάστευση. Μαζί λοιπόν να τα συστήσουμε για να προλάβουμε. Ας δούμε πρώτα τους συνεισηγητές που στο πρόγραμμα εργασίας. Η κυρία Μετσόλα και μετά θα δούμε. Α, η κυρία Αγγιγιώμα αντικαθιστά την κυρία Κέγγε. Καλώς. Κύριε Μετσόλα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Είναι η πρώτη συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ που γίνεται μετά από τις φρικτές επιθέσεις στο Παρίσι και επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή αναδρομή ε, για να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία να δείξω την αλληλεγγύη μου στα θύματα αλλά και να, να, επενέσω τις αστυνομικέ αρχές. Εδώ είναι ακόμα μια δοκιμασία για την Ευρώπη και το πώς θα ανταποκριθούμε θα καθορίσει και την ισχύ των βασικών μας αξιών. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτή την πτυχή. Μετά από αυτές τις ε, φρικιαστικές μέρες, το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιτύχουμε αυτές τις, ε, αφήσουμε αυτές τις επιθέσεις να μας επανακαθορίσουν. Οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που ξεφεύγουν από διώξεις, από τρόμο, από θάνατο και η Ευρώπη πρέπει να δώσει το παράδειγμα για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να ε, έχουν ένα μέλλον χωρίς φόβο. Αυτές οι επιθέσεις γίνανε αδιακρίτα από εγκληματίες και δολοφόνους, όχι πρόσφυγες και θα είχαμε λάθος εάν θέλαμε να τους ε, χαρακτηρίσουμε όλους το ίδιο. Όμως θα πρέπει ταυτόχρονα να είμαστε ρεαλιστές, να μην κρύβουμε το κεφάλι μας στην άμμο. Ο κόσμος έχει φόβους που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση των εξωτερικών μας συνόρων θα πρέπει να γίνει σωστά, να ελέγχεται, να είναι σοβαρός και ισχυρός ο έλεγχος, να ξέρουμε ποιοι μπαίνουν, πού πάνε, Πού βρίσκονται και να επιμείνουμε όλα τα κράτη-μέλη να πληρούν τις υποχρεώσεις τους υπό τον Ευρωπαϊκό Νόμο στα εξωτερικά μας σύνορα. Η ασφάλεια των συμπολιτών μας και των ανθρώπων που χρειάζονται προστασία θα πρέπει να είναι εγγυημένη διαφορετικά. Η ιστορία ότι κατά κάποιο τρόπο οι πρόσφυγες αποτελούν το πρόβλημα θα ε, ε, επικρατήσει. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε το έγγραφο εργασίας μας για την εσωτερική και εξωτερική χρηματοδότηση της Ένωσης σε σχέση με τη μετανάστευση. Είναι ένα από τα οχτώ κεφάλαια της έκθεσης και θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Σεσίλια Κέγκε και όλους καθώς και τον Γιάννη Κορά από την EFTD δεν ήταν πολύ εύκολη η ε, διαδικασία καθόλου μάλλον εύκολη να φτιάξουμε αυτό το έγγραφο ε, και, ναι, και ξέχασα και τη Σεσίλια ε, Βίξτρομ από την Σουλελεύθερος όλοι είχαμε αρκετά ε, γιατί διαφορετικά δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα. Ε, θα επιτρέψω του συναδέλφου να μπουν στα θέματά του, αλλά εγώ θέλω να τονίσω κάποια σημεία κλειδιά. Πώ δαπανώνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια όταν πρόκειται για τη μετανάστευση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το εν λόγω θέμα. Το να πετάμε χρήματα φορολογουμένων σε μια πρόκληση χωρί να έχουμε προγραμματίσει κάτι δεν βοηθά να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Απλά δίνεται εντύπωση ότι κάτι κάνουμε χωρί όμω να προχωράμε πραγματικά. Η Επιτροπή μας ε, εξετάζει λοιπόν τη κονδύλια που υπάρχουν διαθέσιμα για τη μετανάστευση. Ε, εσωτερικά πρέπει να είμαστε σε θέση να δούμε ακριβώς τι κάνει, πόσα δαπανά ακριβώς η Ένωση για τη μεταναστευτική πολιτική. Γι' αυτό πάντοτε, πάντοτε θα μπορούσε να είναι πιο διαφανές, διότι δεν είναι διόλου διαφανές για την ώρα. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο, αναγνωρίζουμε ότι οι πόροι της Ένωσης που αφιερώνονται στο χειρισμό της ε, προσφυγικής κρίσης έχουν αυξηθεί κατά 1,7 δις ευρώ το 2015 και 2016 στους προϋπολογισμούς δηλαδή τους σχετικούς και υπογραμμίζουμε ότι η κοινωνία των πολιτών έχει ένα παίξει ρόλο και ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα πρέπει να καταστεί διαθέσιμη. Εξωτερικώ ζητούμε από τα κρατημέλη να συμβάλλουν περισσότερο στον, ε, ε, στο καταπίστευμα για την Αφρική που πρόσφατα δημιουργήθηκε εδώ από την Ευρώπη, αλλά δυστυχώς ε, οι δωρεές δεν πόρα απέχουν από αυτά που χρειάζονται, δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες. Τώρα, δεν θα πρέπει επίσης να κάνουμε πίσω λόγω των πολλαπλών ε, δημοσιονομικών γραμμών και projects. Ε, ο κόσμος μας θέλει να ξέρει πώς δαπανώνται αυτά τα χρήματα. Να δούμε δηλαδή πού πάνε τα χρήματα και η βοήθεια προς τις χώρες. Σε ποιοι τα παίρνουν και πώς δαπανώνται αν δαπανούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε ο κόσμος αυτές τις χώρες να έχει ένα μέλλον για το οποίο να θέλει να μείνει στην χώρα του. Όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια, όχι την ανθρωπιστική, αναγνωρίζουμε ότι αυτή μπορεί να είναι να, ερετή, δηλαδή να βασίζεται σε όρους Μακροπρόθεσμα θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη όθηση στην επιλύση των γεωπολιτικών ε, θεμάτων που επηρεάζουν τη μετανάστευση. Ω προς αυτό καλούμε την Κομισιόν και τα κατημέλη να οικοδομήσουν ε, δυνατότητε στι τρει χώρες και να εργαστούν για να διευκολύνουν τι επενδύσει στην Αφρική, να βελτιώσουν τι ε, ευκαιρίε για παιδεία, αλλά και να ενισχύσουν τα συστήματα ασύλου, να φτιάξουν καλύτερα συστήματα ελέγχου των συνόρων και καλύτερα συστήματα επιβολή. Τέλο του νόμου. Τέλος όμως, φυσικά τα χρήματα είναι σημαντικά, αλλά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ισότιμη και συγκεκριμένη αλληλεγγύη με συγκεκριμένα μέτρα. Δεν μπορούμε να πετάμε χρήματα στο θέμα και να περιμένουμε να λυθεί μόνο του ή να νομίζουμε ότι αρκετά κάναμε επειδή και μόνο αυξήσαμε κάποιου γραμμέ του προπολογισμού. Πρέπει να ασκήσουμε την πίεση προς κάθε κράτο μέλο ώστε και να κάνουν αυτά που χρειάζονται. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρία Ματσόλα. Και τώρα έχουμε την κυρία Γκυγιόμ που θα μιλήσει εξ ονόματος της κυρίας Κέγκε. Ναι, όντω ε, λαμβάνω το λόγο εξ ονόματο τη συναδέλφου Κέγκε που ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι σήμερα παρούσα εδώ. Καταρχήν θέλει να ευχαριστήσει τι ε, σκιώδει που συμμετείχαν εντατικά στη σύνταξη αυτού του εγγράφου εργασία, την κυρία Κοράου και τη κυρία, και την κυρία Μετσόλα. Ε, η βάση κίνησης ήταν πολύ ε, συμπαγής και γι' αυτό οι δύο εισηγητές μπόρεσαν να φτιάξουν ένα νέο κείμενο με την διαμεσολάβηση των δύο μεγάλων ομάδων και της ΓΚΟΕ και της ΑΛΔΕ. Το έγγραφο αυτό είναι το τέταρτο έγγραφο εργασία ε, σε ένα σύνολο 8 που υποβάλλονται εδώ στη βάση μιας έκθεσης ίδιας πρωτοβουλίας για την ανάγκη στρατηγικής για καθολικής στρατηγικής απέναντι στην μετανάστευση. Είναι δύσκολη η ακριβή κωδικοποίηση των ακριβών δωρεών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών στα θέματα μετανάστευση και ασύλου. Προσπαθήσαμε αυτό να το καθορίσουμε ε, για να δούμε και ποιες πολιτικές δραστηριότητες μπορούν και πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Εγώ θα σας πω κάποιες συστάσεις περιλαμβάνοντας στο έγγραφο και που είναι οι πιο σημαντικές για την κυρία Κέγκε και στοχεύουν στην ε, χορήγηση αλλά και στην εφαρμογή των ε, project αλλά και για το μέλλον. Ακόμα και αν στους προπολογισμού του 2015 και του 2016 υπήρξε αύξηση των διαθέσιμων πόρων στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης, το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων προέρχεται από τα χρήματα που υπάρχουν στο πολιτικό πολιεπτές ώστε η Ένωση να δαπανίσει μέσα στο 2016 τα όσα θα έπρεπε να έχει, ε, θα, μπορούσε, θα μπορούσε να δαπανίσει ανάμεσα στο 2016 και το 20. Επίσης, το ΑΜΥΦ θα πρέπει να γίνει απόλυτα σεβαστό στην, από τα κράτη-μέλη και στην εφαρμογή των πολιετών τους εθνικών προγραμμάτων. Οι βελτιώσεις για το ΑΜΥΦ για τους προπολογισμού 15 και 16 δεν συνοδεύτηκαν από την αναθεώρηση γενικά των κονδυλίων. Δεν θέλουμε να εξαντληθεί γρήγορα το Ταμείο ΑΜΥΦ, θα πρέπει να υπάρξει τέτοια αλλαγή, ε, τροποποίηση. Στον τομέα λοιπόν της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει τα σχετικά project να έχουν την προτεραιότητα από πλευράς Κομισιών και κρατών μελών. Επίσης, θέλουμε να έχουμε πιο, ευκο, ε, πιο ευνόητες, ευανάγνωστες πληροφορίες σε σχέση με τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ε, κρατικό επίπεδο. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται για τα ποσά που δίνονται από τα κράτη-μέλη και από την ε, Κομισιόν για την ε, επιχείρηση Σόφια που προηγούμενα είχε το όνομα ένα φόρ. Ε, πρέπει να υπάρχουν μεμονωμένες γραμμές για καθέναν από τους και τέσσερις κοινού στόχους του ΑΜΕΦ. Πρέπει να εξασφαλιστεί καταλληλότερη ε, χρηματοδότηση για τις ερευνητικές δραστηριότητες και για τις ε, επιχειρήσεις βοήθειας, την επανεγκατάσταση, την εξασφάλιση της πρόσβασης της κοινωνικής υπηρεσίας για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Ενθαρρύνονται επίσης αυτό το κείμενο ε, τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν χρησιμοποιώντα τα ευρωπαϊκά κονδύλια στο μέτρο του δυνατού, χρηματοδοτώντα τι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών που δραστηριοποιούνται στου προαναφερθέντε τομεί. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ ε, θα πρέπει να υπάρξει σημαντική αύξηση των ε, σχετικών κονδυλίων, ειδικά αυτών προορίζονται για το ΑΜΙΦ. Η ε, Κομισιόν επίσης προτείνει η ε, ΤΕΠ να προσφέρει ειδικές, ε, ειδικούς όρους για τα προγράμματα που αφορούν τους μετανάστες που έχουν πρόσφατα έρθει στα κρατημέλη. Για την επιστροφή των μεταναστών θα πρέπει τα κρατημέλη να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με το διαδικαστικό και θεμελιώδες δίκαιο, μάλλον για τα δικαιώματα των εν λόγω ανθρώπων, για τα hot spots που έχουν θεσπιστεί σε κάποια κρατημέλη πρέπει να επιμένουμε ότι οι ΜΚΟ δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται στον έλεγχο αυτών των hot spots για να μας μπορούν να μας ενημερώνουν αν υπάρχουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή διαδικαστικών ε, ε, προβλήματα που υπάρχουν εκεί. Το υπόλοιπο κείμενο είναι στα αγγλικά. Ε, και μετά πάλι στα Χρειάζονται επιπλέον επενδύσεις για να αναπτυχθούν μόνιμες οδοί ε, μετανάστευση όπως μέσα στη στρατηγική 2020. Χρειάζεται ε, έλεγχος των χρημάτων που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μια ασυνέπεια ανάμεσα στα εσωτερικά και τα εξωτερικά κονδύλια, καθώς και ανάγκη για βελτίωση του συντονισμού ανάμεσα στη χρηματοδότηση των πολιτικών μετανάστευσης, ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Σπινέλη έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τις συγκίτριες, ε, την ε, κυρία Κοράου, το προσωπικό μας για την εξαίρετη συνεργασία. Κάποια στη σημεία όμως τα οποία με ενδιαφέραν πολύ δεν βλέπω να έχουν περιληφθεί στην τελική έκδοση, όπως, σε παράδειγμα τη για την ιδιωτικοποίηση των κέντρων υποδοχή, ε, ένα από τους λόγους που οδήγησαν στο σκάνδαλο μαφία στην πρωτεύουσα, στην Ιταλία ή τα κέντρα κατά, καταγραφής ε, και υποδοχής των ετούντων το άσυλο με πολλά προβλήματα που διαπιστώνονται από τις μαρτυρίες. Η αιρεσιμότητα που θα ήθελα να εγγράφεται για βοήθεια προς ε, χώρες ε, μέσα στη διαδικασία του, καρτούμ, του χαρτούμ. Ιδιαίτερα θετικό βρίσκω το να αναφέρεται μία ανάγκη για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και δίωξη των εγκληματιών γραμμές επίσης στον προϋπολογισμό σε σχέση με το Ταμείο Άσυλο, Μετανάστευση, Ενσωμάτωση με διαφορετικούς πόρους και χωριστούς πόρους για, την, ε, για το άσυλο, τη μετανάστευση, την επαναπροώθηση και την αλληλεγγύη μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών. Τρίτον, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί να εμπλακούν ε, κατά μεγάλο βαθμό οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, και να ε, συμμεριστούν και τον έλεγχο και τις ευθύνες ε, στη διαχείριση των κονδυλίων. Άρα χρειάζονται μηχανισμοί παρακολούθησης και αξιολόγηση όχι μόνο εκ των υστερών αλλά και κατά τη διάρκεια εξέλιξης των προγραμμάτων ώστε να παριθεύεται ότι τηρούνται οι στόχοι. Αυτά λένε τα θετικά της εκθέσεως και εν τέλει βλέπω ότι υπάρχει ένα αίτημα για σταθερή χρηματοδότηση και υποστήριξη από την Ένωση και των διεθνών οργανώσεων που είναι παρούσες στους ε, χώρους όπου εμφανίζονται τα οι ανάγκες για τους πρόσφυγες και μετανάστες και βέβαια σύστημα άμεσης πριμδότησης, για τις πιο μικρές δομές και μη κυβερνητικέ οργανώσεις κυρίως που θα έχουν ανάγκη για πρόσβαση πιο γρήγορη στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ζητώ συγγνώμη ε, από τους συνοδέλφους που θα χρειαστεί να, να αποχωρήσω πολύ σύντομα γιατί έχω μία συνεδρίαση που δεν μπορώ με κανένα τρόπο να αποφύγω. Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ και πάλι συγγνώμη που θα φύγω. Κοράω. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την συνάδελφο Σπινέλη και το... όπως η κυρία Σπινέλη και το προσωπικό μας και όλους τους συναδέλφους ε, και βέβαια την κυρία Μετσόλα και την κυρία Κέντζε συνεισηγήτριες είναι προϊόν συμβιβασμού βέβαια η έκθεση που εξετάζουμε. Αυτός ήταν και ο στόχος τον οποίο είχαμε ορίσει ξεκινώντας να υπάρξει πολιτική συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Άρα προφανώς και κάπως υποβαθμίστηκαν οι προσδοκίες μας. Όντας Ιταλός και Σικελός συγκεκριμένα, εγώ θα είχα ακόμη πιο άτεγκτη στάση ως προς σημεία, αλλά όπως λέω, έστω προκειμένου να εξευρεθεί μια ε, εγκάρσια συνένεση μεταξύ των πάντων για να προχωρήσουμε περισσότερο, ας το δεχθούμε. Βεβαίως πολύ συχνά είδαμε ε, το οργανωμένο έγκλημα και πιο συγκεκριμένα η μαφία να ε, διαπλέκονται με την πολιτική για να καθοδηγήσουν μεταναστευτικές ροές και να μετατρέπουν τις μεταναστευτικές ροές σε επιχείρηση επικερδή. Ε, όταν μιλούμε για κονδύλια πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δεν είναι απεριόριστα, άρα πρέπει να κατανέμονται κατά τρόπο ορθό και με βάση τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλογικά και προς τις ανάγκες των κρατών μελών και λαμβάνοντας υπόψη διάφορες ε, πτυχές των αναγκών και της κατεπίγουσας κατάστασης στην Ένωση η διάσωση στη θάλασσα, οι επαρκείς και σωστές δομές υποδοχής, η επαναεγκατάσταση στις κοινωνίες μας, η κοινωνία των πολιτών που μπορεί να στηρίξει τους πρόσφυγες και μετανάστες είναι διάφορες πτυχές, ιδιαίτερα σημαντικές σε μια ορθή πολιτική μετανάστευση και δεν μπορούν να θυσιαστούν στον βωμό της απλής εποπτείας των συνόρων. Ιδιαίτερα πρέπει να μιλήσουμε για την πρόληψη και την κύρωση βάρος των καταχρήσεων ε, ιδιαίτερα όσον αφορά κονδύλια που χρηματοδοτούν ε, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και για τα οποία δεν υπάρχουν πάντα δυνατότητες για επαλήθευση και ενημέρωση. Η διαφάνεια λοιπόν απαιτείται μέσα σε ένα πλέγμα το οποίο είναι αρκετά περίπλοκο και δεν επιτρέπεται η δημοκρατική λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, η αδιαφάνεια λοιπόν μετατρέπει την επιχείρηση διακίνησης μεταναστών και προσφύγων σε μια επικερδή επιχείρηση οδηγεί σε μια πελατειακή σχέση μεταξύ δικτύων και ε, δικτύων εγκληματιών και μεταναστών ή προσφύγων όπως αποδείχθηκε και από το σκάνδαλο Μάφια Καπιτάλη, η μαφία στην πρωτεύουσα δηλαδή Αυτά όλα είναι στόχοι που πρέπει να καταπολεμηθούν, που καταγράφονται στην έκθεση τώρα θέλουμε να υπογραμμίσουμε και πιστεύω ότι πρέπει ε, τα κονδύλια να αξιοποιούνται κατά τρόπο ορθολογικό για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων με βάση τις ανάγκες των κρατών μελών και των τρίτων κρατών, να προάγουν έναν τρόπο διαχείρισης, παρακολούθησης, εποπτείας ε, και διαφανούς ελέγχου της διαχείρισης των κονδυλίων, να επενδύουν σε νόμιμα πάνω απ' όλα μέσα ε, εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους μετανάστες και πρόσφυγες και προγράμματα χρηματοδότησης διαφορών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα χρειαστούν προκειμένου να ε, στηριχθούν και οι διάφοροι φορείς από την κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ θερμά. Uh, και τώρα ζητώ όσους ε, θέλουν να πάρουν το λόγο. Η κυρία Γκόμες, σύντομα. Θα ήθελα να πω ότι δεν νομίζω πως ε, η διαδικασία του Χαρτούμ μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα σύστημα ανάθεσης εξωτερικούς ε, συνεργάτες ή υπεργολάβους ε, πραγμάτων που εμείς δεν αντέχουμε να επιτελέσουμε. Δεν γίνεται αυτό. Και δεύτερον, θέλω να πω ότι χρειάζεται περισσότερη συνοχή και επικοινωνία, μια διαδραστική θα λέγαμε σχέση μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής διάστασης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Εν προκειμένου λοιπόν θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία, όπως την περιέγραψε ο Επίτροπος Χάν και η υπατή εκπρόσωπος ε, Μογκερίνη, μπορεί να είναι σημαντική και πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στην έκθεση. Να αντικατοπτρίσετε λοιπόν αυτή η διαδραστική σχέση. Βλέπουμε μεγάλη απουσία συντονισμού. Απαράδεκτη απουσία συντονισμού, δεν μπορεί να συνεχιστεί. γιατί θα συνεχίσουν να καταφθάνουν μετανάστες και πρόσφυγες και μέχρι ότου ή εφόσον ή εάν δεν ορίσουμε νόμιμους τρόπους μετανάστευσης και εισόδου δεν θα απαλλαγούμε από το πρόβλημα. Και βεβαίως ε, δεν υπάρχει τρόπος να αποτρέψουμε την άφηξη Είχαμε πρόσφατα επικοινωνία με μη κυβερνητικέ οργανώσει που προσφέρουν αρρωγή στου ε, πρόσφυγε που βρίσκονται στην Τουρκία αλλά και σε άλλε χώρε τη περιοχή και μία από τι ε, περιπτώσει που μου περιγράφηκε ήταν αυτή του Ιράκ όπου μεταξύ της ΕΚΟ και της, μακροπρόθεσμης, ε, της υπηρεσίας για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη δεν υπάρχει στονισμός. Δηλαδή δεν προσφέρονται σχολεία, γιατί αυτή θα ήταν αρμόδιοι για τα σχολεία. Δεν προσφέρονται σχολεία στους καταβλισμούς των προσφύγων στο, Ιράκ ε, για τους εσωτερικά εκτοπιστέντες, ε, για αυτούς που φεύγουν για να γλιτώσουν από το Ίκυρ. Δεν υπάρχουν σχολεία για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν καν μέλλον για τα παιδιά τους. Και δεν θα έχουν τα παιδιά τους μέλλον εάν δεν τους δοθεί σχολική εκπαίδευση. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν αυτή η απουσία διασύνδεσης και επικοινωνίας να συνεχιστεί. Η κυρία Μετσόλα, η κυρία Κέγκε, τι οποίε και συγχαίρω για την πολύ καλή δουλειά τους και συμφωνώ μαζί τους, είμαι βέβαιο ότι θα το αναλάβουν. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να πω ότι πήγα στα Δυτικά Βαλκάνια με την QNGL, έκανα μια αποστολή και ε, πήγαμε σε πολλά κέντρα ε, διέλευσης καλά. Πήγαμε στα Δυτικά Βαλκάνια και περάσαμε σε, πολλά, ε, σε πολλούς καταβλισμούς διέλευσης στη Ποτροβιάνα στα σύνορα Βουλγαρίας, Σερβίας. Ήταν ένα από αυτά τα κέντρα και ε, κάποιοι πρόσφυγες ε, είχαν ξυλοκοπηθεί από τις ε, αρχές, τους είχαν κλέψει. Τους είχαν δαγκώσει τα σκυλιά των συνοριοφυλάκων και αναρωτιέμαι Υπάρχει καμιά ε, δυνατότητα έρευνας από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ή αναστολής ε, της χρηματοδότησης όταν υπάρχουν καταχρήσει από πλευράς της αστυνομίας όπως η συγκεκριμένη περίπτωση. Ευχαριστούμε και συγγνώμη για το πρόβλημα με τη διερμηνία. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μετσόλα, εφόσον δεν θέλει κάποιος άλλος το λόγο, για να περάσουμε άμεσως στο επόμενο σημείο για την ε, αντιπροσωπεία στην Τίνιδα. Παρακαλώ. Um, well, no. Ευχαριστώ. Σημείωσα όλα τα σχόλια που ε, ακούσαμε. Θα ήθελα να συνεχίσω τις προσπάθειες που κάνουμε για να καταλήξουμε συμβαστικές λύσεις με τις πολιτικές ομάδες. Για την πολιτική γειτονία καταλαβαίνω αυτά που είπατε κυρία Γκόμες και θα τα πάρω ε, ε, υπόψη μου στον μέλλον. Σίγουρα ε, στην τελική έκθεση θα συμπεριλάβουμε αυτά τα σχόλια και ευχαριστούμε για την υπόδειξη. Για την ίδια έκθεση, την ίδια έκθεση για την, την νομίζω ότι δεν χρειάζεται να προσθέσω εγώ ε, κάτι. Ε, ήταν εξαιρετική η αντιπροσωπεία, η Σεσίλ Κέγγε και υποφαινόμενη υποφαινόμενοι. Γηθήκαμε της πέντε μελών της Επιτροπής και ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένο το πρόγραμμα. Ευχαριστώ τη γραμματεία παρεμπιπτόντως. Είχαμε ξεκαθαρίσει πως θέλαμε να ε, υπερβούμε αυτά που έκαναν προηγούμενε αντιπροσωπείε σε, σε βορειοαφρικανικές χώρες, δηλαδή να συναντούμαστε με εκπροσώπου των κυβερνήσεων και να ακούμε μόνο τη μία πλευρά, ας, το πούμε, ας πούμε την αλήθεια. Ε, και μετά την απονομή ε, του βραβείου Νόμπελ συναντήκαμε μαζί τους ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εφημερίδες, ε, ήρθανε όλοι να μας πούν πώς είναι η πραγματικότητα επί τόπου. Η... Τα δύναμα ε, σημεία της ε, ε, σχετίζονται με την ε, Λιβύη, ειδικά στις μεθοριακές περιοχές. Υπάρχουν προβλήματα διότι προκύπτουν επιθέσεις ή μπαίνουν ένοπλοι πετράπει μία επίθεση τις τελευταίες ημέρες, ακόμη μία, όμως ε, δεν υπάρχει δυνατότητα δράσης ε, διπλωματική οδού ε, και αναπτύσσονται ισλαμιστικοί πυρήνες από πλευράς Ίσης και Μποκοχαράμ στο, στη βόρεια την Ισία. Και ε, αυτό είναι άμεση ε, απόρρια της κατάστασης ε, στην ε, Λιβύη. Αντίθετα, η συνεργασία με την Αλγερία από την άλλη πλευρά είναι καλή και μετά τις επιθέσεις της ΣΟΥΣ δέχτηκαν αρρωγή την νησιακές αρχές Πήγαμε στο κέντρο υποδοχής ή κράτησης, νοτιασί, ας το πούμε κράτησης, ένας υπήρχε μόνο μέσα στο κέντρο και μας δώσαν την εντύπωση ότι όλα πηγαίνουν καλά. Προβληματίστηκα για το τι σημαίνει στην πραγματικότητα. Πού είναι οι άνθρωποι αυτοί Πού είναι αυτοί που διαμένουν εκεί παράνομα. Αν δεν είναι στα κέντρα κράτησης υποθέτω είναι σε φρονιστικά ιδρύματα. Παρόλα αυτά, χάρη στη συνάντηση αυτή καταφέραμε να διαμορφώσουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα που γεωγραφικά είναι ε, πολύ κοντά στην Ευρώπη, γιατί μιλήσαμε και για τη Σικελία προηγουμένως. Καλό θα ήταν να οργανώσουμε και άλλες συναντήσεις γιατί οι δύο γειτονικέ χώρες ε, παλεύουν ε, με, τα, με τις μεταναστευτικές ροές δεν ανθεί πλέον ε, η ριζοσπαστικοποίηση και συνεχίσετε παρόλα αυτά ε, η διακίνηση ανθρώπων. Συναντηθήκαμε επίσης με πολλούς εκπροσώπους των προξενείων και των ε, πρεσβειών επιτόπου κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους ρωτήσαμε τελικά η την Ισία είναι χώρα διέλευσης ή τελικός προορισμός. Ένας εκπρόσωπος μας είπε ότι οι περισσότεροι που ζητούν θεώρηση εισόδου είναι την ίση και θέλουν να έρθουν για να δουλέψουν στην Ένωση αντίθετα με αυτό που μας είπε ο υπουργό Εσωτερικών, που παρουσίασε μια εικόνα ε, θετική. Όσοι είναι από τα 18 μέχρι τα 35, κυρίως οι άντρες, θέλουν να μπουν στην Ευρώπη για να εργαστούν ή να σπουδάσουν ανάλογα με την κατάστασή τους. Αυτά τα στοιχεία έχουμε εμείς. Ευχαριστούμε, Ρομπέρτα. Ο κύριος Κοράου ε, αντικαθιστά την κυρία Κένια. Ευχαριστώ. Μιλώ εκ μέρου και τη κυρία Κένγκε, αλλά και προσωπικώ, καθώ είμαι μέλο αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την Ισία. Συμφωνώ με τα όσα μα περιέγραψε η Ρομπέρτα Μετσόλα και ευχαριστώ ιδιαίτερα στη Γραμματεία για την πολύ καλή δουλειά που έκανε αυτές τις δύο ημέρες όπου πρακτικά δεν είχαμε ούτε ένα λεπτό να, για, ούτε μια λεπτό για μια ανάσα. Είχαμε διαρκείς συναντήσεις, μεταβάσεις από το ένα μέρος στο άλλο, από το πρωί στο βράδυ. Πιο γεμάτο πρόγραμμα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε στο χρονικό αυτό διάστημα που έχουμε θέση μας. Αυτό που θα μπορούσα να προσθέσω στα συμπεράσματα και την περιγραφή που ακούσαμε. από τις συζητήσεις, τις επαφές που είχαμε με την κοινωνία των πολιτών και τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, της Βουλής, των θεσμών της Τινησίας αντελήφθημεν ότι έχει πολύ μεγάλη έμφαση δώσει στην προτεραιότητα της ασφάλειας η κυβέρνηση και την ανάπτυξη μιας πολιτικής μετανάστευσης ε, περιεκτικής και αποτελεσματικής. Έτσι λοιπόν, όπως ε, αντιλαμβανόμαστε από αυτές τις ε, συζητήσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις αρχές της Τινησίας να αναγνωριστεί ότι δεν είναι πια χώρα διέλευσης αλλά χώρα προορισμού η Τινησία. Άρα χρειάζεται μια οργανική νομοθεσία για την μετανάστευση. Η χώρα δεν έχει νομοθεσία για το άσυλο και άρα χρειάζεται το ταχύτερο δυνατό να προβλεφθεί αυτό και επίσης φαίνεται να μην κατέστη απόλυτα σαφές ε, στις επαφές μας με τους βουλευτές ε, το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναμένεται να υιοθετηθεί αυτή η νέα νομοθεσία για το άσυλο. Και βέβαια το καθεστώς, το νομικό καθεστώς των μεταναστών έχει ακόμα, μένει ακόμα να διευκρινιστεί. Το ζήτημα της νομιμοποίησης που απουσιάζει αυτή τη στιγμή και έτσι αυτομάτως ε, είναι διαπράττουν αδίκημα όποιοι περνούν τα σύνορα γιατί δεν έχουν νόμιμη είσοδο και άρα πρέπει να πληρώνουν καθημερινό πρόστιμο 20 διναρίων για κάθε μέρα που βρίσκονται αλλά δεν είναι σε θέση και να βγουν από τη χώρα γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το πρόστιμο προκειμένου να τους επιτραπεί να διασχίσουν και πάλι τα σύνορα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα νομικής βεβαιότητας ή καλύτερα νομικής αβεβαιότητας και δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ κύριε Κοράο. Κυρία Γκόμες έχει στήσει το λόγο. Για τους συναδέλφους που ήταν σε αυτή την αποστολή θέλω να ρωτήσω το εξή. Από ό,τι γνωρίζω σε τέτοιες ε, αποστολές πάντα φροντίζουμε να έχουμε επικοινωνία με την αντιπολίτευση και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των επισκέψεών μας και πολύ σωστά. Και θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερως τα λόγια της κυρίας Μετσόλα για τις συνέπειες της κατάστασης στη Λιβύη, όχι μόνο για την ασφάλεια της Τινησίας, αλλά για την ασφάλεια όλων μας. Και πάλι εδώ τα κράτη-μέλη, κατά τρόπο γελίο, παραγνωρίζουν τη σοβαρότητα του προβλήματο. Μπορεί κάποια που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να κάνουν περισσότερα πράγματα, αλλά τα περισσότερα παραγνωρίζουν τη σοβαρότητα τη κατάσταση, γιατί η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι το Ισλαμικό κράτο κατέχει εδάφη στη Λιβύη, ελέγχει ήδη εδάφη στη Λιβύη, στη Σύρτη συγκεκριμένα. Στην Τόρνα είχαν πάρει τον έλεγχο αλλά τους έδιωξαν οι πολίτες και τώρα είναι στη Σύρτη, δεν το λέει κανείς και βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να αποσιωπούν τον διαντιπροσώπου πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το No Man's Land, σε αυτό το άντρο του Ίκυλ, το κατασφαλές καταφύγιο για το Ίκυλ και το ρόλο άλλων δυνάμεων και δι Τουρκίας, Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας, Εμμυράτων, ε, Τουρκίας, Κατάρ αφενός, αλλά και Σαουδικής Αραβίας, Εμμυράτων, Αιγύπτου, Αφετέρου, για την κατάσταση αυτή που θα μας οδηγήσει σε μια κατάσταση ακόμα χειρότερη από αυτή που βλέπουμε στη Συρία και το Ιράκ. Αυτά για να μην μου πείτε ότι δεν σας θα είπα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκόμες και αγαπητοί συνάδελφοι για τη συνεργασία. Έχουμε προβλέψει προσεχή συζήτηση για την έκθεση ιδέας πρωτοβουλίας στις 10 Δεκεμβρίου και έτσι το μόνο που μου μένει είναι να ανακοινώσω την προσεχή συνεδρίαση όπως σας ανακοίνωσα εξ αρχής Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 7 με 8 το βράδυ με ψηφοφορίες και γι' αυτό σας παρακαλώ να μην λησμονήσετε τις ε, κάρτες σας για την ψηφοφορία. Κατά τα άλλα, 30 Νοεμβρίου, 1η Δεκεμβρίου, τακτική μας συνεδρίαση και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, την προσοχή σας και τη συνεργασία σας σήμερα, γιατί είχαμε πολύ και δύσκολη δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ και το Σαββατοκύριακο.